Καλημέρα σας, καλησπέρα σας μάλλον κυρίες και κύριοι. Σας καλωσορίζω στην απογευματινή συνεδρίαση αυτή της Επιτροπής ε, Δικαιωμάτων των Γυναικών και Ισότητας των Φύλων. Πολύ ενδιαφέρον προαναγγέλλεται το απόγευμα γιατί θα έχουμε την ευκαιρία να ακούσουμε τις προτεραιότητες της Πολωνικής Προεδρίας στην Ευρωπαϊκή Ένωση και μετά έχουμε πολύ σημαντικές ψηφοφορίες να κάνουμε. Καλώ ήρθατε και πάλι λοιπόν στη συνεδρίαση τη Επιτροπή Δικαιωμάτων των Γυναικών και Ισότητα των Φύλων. Πρώτο σημείο τη ημερήσια διάταξη φυσικά είναι η έγκριση του σχεδίου ημερήσια διάταξη. Και να σα επισημάνω μερικές αλλαγέ που γίνονται στην ημερήσια διάταξη. πρώτη πρόταση αλλαγή αφορά την ψηφοφορία στο σημείο 8 της ημερήσιας διάταξης την έκθεση δηλαδή της κυρίας ε, Σξιδλεύσκα. Το ψηφίο 8 θα είναι το πρώτο θέμα που θα ψηφίσουμε το απόγευμα. Δηλαδή, μετά το 5 της ανακοινώσης Προέδρου θα ψηφίσουμε καταρχήν το σημείο 8 πρώτο. Δεύτερη αλλαγή. Η κυρία Ζαμπόρσκα έχει δύο εκθέσει στην ημερήσια διάταξη τα σημεία 12 και 14. Ζήτησε να συζητήσουμε σήμερα το απόγευμα το 12, αμέσω μετά το πέρας των ψηφοφοριών. Και αν μας περισσέψει χρόνος, θα περάσουμε και στο σημείο 14. Αυτό θα εξαρτηθεί φυσικά από το πόσο χρόνο θα έχουμε στη διάθεσή μας. Είναι θέμα χρόνου. Ευελπιστούμε πάντως ότι στη διάρκεια του απογεύματος θα καταφέρουμε να διεκπαιρεώσουμε και το 12 και το 14. Σε ό,τι αφορά το σημείο 11, το αναβάλουμε για αύριο το πρωί που θα είναι το πρώτο σημείο στην αυριανή ημερήσια διάταξη. Αυτές λοιπόν οι προτάσεις ε, για αλλαγή της ημερήσιας διάταξης και αν δεν έχετε αντιρρήσεις προτείνω να την εγκρίνουμε. Δεν βλέπω αντιρρήσεις. Πολύ ωραία. Εγκρίνεται η ημερήσια διάταξη και περνάμε στο σημείο 2 τις ανακοινώσεις της Προέδρου. Δύο είναι οι ανακοινώσεις μου και παρακαλώ να τις σημειώσετε. 31 Αυγούστου, καταρχήν, στις 31 Αυγούστου η Επιτροπή Πολιτικών Ελευθεριών θα συνεδριάσει με τους συντονιστές για να εξετάσει το θέμα της καταπολέμησης του εμπορίου, σωματεμπορία, εμπορία ανθρωπίνων όντων. Σημειώστε λοιπόν στο πρόγραμμά σα τη 31 Αυγούστου συνεδρίαση με τους συντονιστέ στην Επιτροπή Πολιτικών Ελευθεριών. Αυτή είναι η αρχική πρόβλεψη, ο αρχικός προγραμματισμός. Θα σας μοιράσουμε την αναλυτική μερίσια διάταξη όταν καθοριστεί. Δεύτερη ανακοίνωση Πρόεδρου. Στην επόμενη μας συνεδρίαση, που θα είναι το Σεπτέμβριο στο Στρασβούργο, 15 Σεπτεμβρίου για την ακρίβεια, 9 με 10 και μισή, 15 Σεπτεμβρίου στο Στρασβούργο, προβλέπεται έκτακτη συνεδρίαση της Επιτροπής μας ε, και την περιλάβαμε στο πρόγραμμα γιατί θα χρειαστεί να ψηφίσουμε. Μία έκτακτη συνεδρίαση λοιπόν της Επιτροπής μας στις 15 Σεπτεμβρίου, 9 με 10.30 το πρωί, στο Στρασβούργο. Περνάμε τώρα στο σημείο 3, την έγκριση των πρακτικών. Των πρακτικών της συνεδρίασης της 9ης Μαΐου του 2011. Θα βρείτε στο δοσιέ σας τα πρακτικά και αν δεν υπάρχουν αντιρρήσεις για τα πρακτικά και δεν υποβληθούν μέχρι το πέρας συνεδρίασης, θα θεωρηθούν ως εγκεκριμένα. Ας προχωρήσουμε λοιπόν τώρα στο θέμα 4. Πρέπει να σας πω ότι είμαι ενθουσιασμένη γιατί βλέπω ότι η Επιτροπή μας σήμερα το απόγευμα θα έχει την ευκαιρία να ακούσει περισσότερες λεπτομέρειες σχετικά με τις προτεραιότητες της Πολωνικής Προεδρίας και θα έχει την ευκαιρία επίσης να θέσει ερωτήσεις ή στην Προεδρία και θα έχουμε και τη δυνατότητα μια συζήτησης με την Προεδρία. Χαίρομαι λοιπόν να καλωσορίσω την ε, κυρία Γιολάντα Φέντακ, Υπουργό Εργασίας και Κοινωνικής Πολιτικής και επιπλέον θέλω συγχρόνως να καλωσορίσω και την κυρία Ελσβέτα Ραντζιέσκα, πληρεξούσια της πολωνικής κυβέρνησης για την ίση μεταχείριση. Σας καλωσορίζω, σας καλωσορίζω στο Κοινοβούλιο και στην Επιτροπή Δικαιωμάτων των Γυναικών και Ισότητας των Φύλων και ε, προσλέπουμε σε μία ευχάριστη ε, συζήτηση. Στη συνέχεια θέλω να δώσω το λόγο πρώτα στην κυρία Φέντα, η οποία θα μας κάνει την παρουσίαση. Κυρία Υπουργέ, έχετε το λόγο. Κυρία Πρόεδρε, κυρίες και κύριοι. Αισθάνομαι ιδιαίτερη χαρά για την ευκαιρία που έχω να παρουσιάσω στην Επιτροπή σας τις προτεραιότητες της Πολωνικής Προεδρίας για την ισότητα των δύο φύλων, την ίση μεταχείριση στην πρόσληψη και στην κοινωνική πολιτική. Το γενικό μήνυμα των προτεραιοτήτων μας είναι περισσότερη και πιο αλληλέγγυη Ευρώπη. Στην Πολωνία τα τελευταία χρόνια υιοθετήθηκαν πολλές νομικές διατάξεις που επηρεάζουν ουσιαστικά το θέμα της ισότητας των δύο φύλων. Από το 2008 θεσπίσαμε διατάξεις της πολιτικής για την οικογένεια. Το 2010 αναθεωρήθηκε ο νόμος για την ενδοοικογενειακή βία και επίσης εγκρίθηκε ο νόμος για την ίση μεταχείριση. Ενώ το 2011, φέτος δηλαδή, τέθηκαν σε ισχύ δύο νόμοι. Ο νόμος για τις ποσοστώσεις ε, στους καταλόγους, στις λίστες των κομμάτων, καθώς και ο νόμος για τους βρεφονιμπιακούς σταθμούς. Μία από τις ε, πρωταρχικές προτεραιότητες της Πολωνικής Προεδρίας σε θέματα απασχόλησης και κοινωνικών δικαιωμάτων είναι η, η αλληλεγγύη μεταξύ των γενεών σε ό,τι αφορά το δημογραφικό μέλλον της Ευρώπης. Και Πολλές ε, δραστηριότητες θα έχουν στόχο το να δώσουμε νέα όθηση για την ε, ενεργοποίηση της ε, επαγγελματική δραστηριότητας και την ανέβρεση λύσεων που θα διευκολύνουν τον συνδυασμό του επαγγελματικού με τον οικογενειακό βίο και για τις γυναίκες και για τους άντρες. Η Πολωνία κατά τη διάρκεια της προεδρίας της στο Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης θα δώσει ιδιαίτερη προσοχή στα εξής θέματα στην ενίσχυση της συμμετοχής των γυναικών στην αγορά εργασίας και στις διάφορες διαδικασίες λήψης αποφάσεων, κοινωνικών και πολιτικών, τη συμφιλίωση του επαγγελματικού και του οικογενειακού ρόλου των ανδρών και των γυναικών και επίσης ε, την καταπολέμηση της ενδοοικογενειακής βίας. Στα πλαίσια των προγραμματισμένων προτεραιοτήτων Τη Πολωνική Προεδρία για την ε, αλληλεγγύη μεταξύ των γυναικών στο πλευρό του δημογραφικού, δημογραφικού τη Ευρώπη, προβλέπουμε να ε, προωθήσουμε την ενίσχυση τη ε, απασχόληση των ανδρών και γυναικών, την δυνατότητα επαγγελματική καλύτερη δραστηριοποίηση των γυναικών σε κάθε βαθμίδα ιδιοδρομία, να ε, διευκολύνουμε την αναπρόσωπηση γυναικών μετά την ε, άδεια μητρότητα ή γονική άδεια και την επαναφορά του στην αγορά εργασία μετά το 50ο έτος ηλικία ή μετά από μακροχρόνια ανεργία. Όλε αυτέ οι δραστηριότητε που θα ε, αναλυφθούν από το Υπουργείο μας θα δρομολογηθούν μέσω διαφόρων προγραμμάτων όπως την κοινωνική και οικονομική δραστηριοποίηση των γυναικών σε τοπικό και περιφερειακό επίπεδο, το συνδυασμό του επαγγελματικού και οικογενειακού ρόλου ανδρών και γυναικών και το gender mainstreaming ως τρόπο και εργαλείο αλλαγών στην αγορά εργασία. Έχουμε σχεδιάσει και άλλες δραστηριότητες για να ενισχύσουμε την ενεργό συμμετοχή των γυναικών στον κοινωνικό και δημόσιο βίο. Και από τα σημαντικότερα προγράμματα του Υπουργείου μας στον τομέα αυτό είναι η συνδιοργάνωση του Συνεδρίου των Γυναικών. Η φετινή οργάνωση, που θα είναι η τρίτη οργάνωση αυτού του Ευρωπαϊκού Συνεδρίου, θέλουμε να δώσουμε έναν διακρατικό, διεθνή χαρακτήρα και μάλιστα αυτό θα είναι μια σημαντική δραστηριότητα του Υπουργείου μας κατά τη διάρκεια της Πολωνικής Προεδρίας. Πρόκειται για μια εκδήλωση που θα διοργανωθεί στη Βαρσοβία 17 και 18 Σεπτεμβρίου και μάλιστα σας προσκαλούμε θερμά σε αυτή τη διοργάνωση του Ευρωπαϊκού Συνεδρίου Γυναικών που θα γίνει υπό την αιγύδα του Πρόεδρου μας. Θα συζητήσουμε πολύ σημαντικά θέματα για τις γυναίκες. Γι' αυτό θα ήθελα να προσκαλέσω και εσάς και τους βοηθούς σας στο συνέδριο αυτό. Η φετινή λοιπόν οργάνωση του συνεδρίου θα έχει ευρωπαϊκό, πανευρωπαϊκό χαρακτήρα θα οργανωθεί, όπως σας είπα, υπό την αιγίδα της Πολωνικής Προεδρίας. Θα διοργανώσουμε πάνελ συζητήσεων και μια στρογγυλή τράπεζα, στην οποία θα συμμετέχουν γυναίκες υπουργοί για θέματα ισότητας. Θα συμμετέχουν λοιπόν επίσης εμπειρογνώμονες και εκεί θα γίνεται ανταλλαγή απόψεων με θέμα τις διαφορές στην στις αμοιβέ για τους άνδρες και τις γυναίκες. Θα εξεταστούν ε, εύρυθοι μηχανισμοί του συνδυασμού του επαγγελματικού και οικογενειακού ρόλου και το θέμα της ενίσχυσης της συμμετοχής των γυναικών στα διοικητικά συμβούλια των επιχειρήσεων. Στη διάρκεια της Πολωνικής Προεδρίας, ιδιαίτερη έμφαση δίνουμε στην πρόθεση κάποιων μηχανισμών που θα διευκολύνουν τη συμμετοχή των γυναικών στην αγορά εργασίας προγραμματίσαμε άτυπο Συμβούλιο Υπουργών Ισότητας Φίλων και Οικογένειας, καθώς και μία διάσκεψη εμπειρογνωμόνων με θέμα τους μηχανισμούς συμφιλίωσης του επαγγελματικού και οικογενειακού ρόλου για τις γυναίκες και τους άντρες και μία ευκαιρία για ενεργό συμμετοχή στην αγορά εργασίας. Και οι δύο αυτές εκδηλώσεις έχουν προγραμματιστεί για φέτος τον Οκτώβριο στην Κρακοβία και φυσικά και για τις δύο διασκέψεις ε, προσκαλούμε τους βουλευτές, τα μέλη της ε, δικής σας επιτροπής. Θέλουμε να κάνουμε μια επισκόπηση και τον πρόοδων που έχουμε κάνει στα θέματα ισότητας φύλων και να τοπίσουμε τις βασικές προκλήσεις που αντιμετωπίζουν τα κράτη-μέλη. Η ανταλλαγή βέλτιση των πρακτικών ε, και η εξέταση εύρυθμων μηχανισμών προκειμένου να προωθήσουμε και να ενισχύσουμε τις προσπάθειές μας για να εξαλείψουμε τις διαφορές και να συγκεντρώσουμε ε, πληροφορίες για τις επιβλαβείς πρακτικές προκειμένου να θεσπίσουμε τις διατάξεις για την κατάργηση αυτών των επιβλαβών πρακτικών. Στη διάρκεια της διάσκεψης αυτής και από τα Υπουργεία της Δανίας και της Κύπρου θα ε, προσυπογράψουμε μία διακήρυξη για το θέμα της ε, ισότητα των φύλων κατά το 18μηνο του Τρίου των Προεδριών. Επίσης, θα χρησιμοποιηθεί αυτό το φόρουμ για την ανταλλαγή βέλτιστων των πρακτικών μεταξύ των κρατών μελών και θα μπορέσουμε να κάνουμε μια επισκόπηση των προόδων που έχουμε σημειώσει σε θέματα ισότητας φύλων και πάλι θα εξετάσουμε τις βασικές ε, προκλήσεις που αντιμετωπίζουν τα κράτη-μέλη και θα προωθήσουμε περαιτέρω προσπάθειες με στόχο την εξάλληψη των διαφορών. Οι, οι, τα μέλη και οι, όσοι θα συμμετέχουν και στην ε, υπουργική διάσκεψη αλλά και στην διάσκεψη των εμπειρογνωμόνων θα λάβουν γνώση και της έκθεσης που εκπονεί το Ευρωπαϊκό Ινστιτούτο Ισότητας Φίλων του Βίλνιους ειδικά μάλιστα κατέθεση της Πολωνικής Προεδρίας. Η έκθεση αυτή θα περιλαμβάνει μία επισκόπηση των ε, διαφόρων δράσεων της πλατφόρμας του Πεκίνου ε, με θέμα κυρίως ε, τις γυναίκες και την οικονομία. Σε ό,τι αφορά παραδείγματα πολωνικών δραστηριοτήτων στον τομέα αυτό και τέτοιου είδους παραδείγματα θα υποβληθούν στις δύο αυτές διασκέψεις που σας ανέφερα. Μάλιστα πρόσφατα ε, εγκρίναμε στην Πολωνία το νόμο για τη φροντίδα των ε, μικρών παιδιών κάτω των τριών ετών. Αυτό τον ε, νόμο τον αποκαλούμε κοινό νόμος για τους βρεφονιπιακούς σταθμούς και προτείνει διαφοροποιημένες μορφές για τη φροντίδα παιδιών ω τριών ετών. Και επίσης παροτρύνει τους εργοδότες να προβλέψουν και εντός ή κοντά στις επιχειρήσεις τους τέτοιους βρεφονιπιακούς σταθμούς. Ο νόμος αυτός για τους βρεφονιπιακούς σταθμούς προσπαθεί να ανταποκριθεί στις προσδοκίες των γονιών που θέλουν να συμφιλιώσουν τον επαγγελματικό και τον οικογενειακό τους ρόλο. Και μάλιστα από τον Ιανουάριο του 2010 ο Πολωνικός Εργατικός Κώδικας προβλέπει τη δυνατότητα χορήγησης επιπλέον άδειας μητρότητας αλλά και άδειας πατρότητας. Αυτά τα στοιχεία θα υποβληθούν ε, ως καλές πρακτικές της Πολωνίας στην διάσκεψη αυτή. Το Μάρτιο του 2011 το Εθνικό Κέντρο ε, Αρμοδιότητας σε συνεργασία με το Υπουργείο μας ε, οργάνωσε στην Πολωνία μια διεθνή διάσκεψη κατά τη διάρκεια της οποίας συμμετείχαν εκπρόσωποι όλων των κρατών μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης και εξετάστηκε το θέμα της καταπολέμησης της ενδοοικογενειακής βίας. Άλλωστε έχουμε και την πρόταση της Ευρωπαϊκής ε, Κοινωνικής Εκστρατείας για την καταπολέμηση της ενδοοικογενειακής βίας με τίτλο «Αγαπώ, δεν χτυπώ». Στη διάρκεια της Πολωνικής Προεδρίας, το Προεδρείο μας ε, θα συμβάλλει ενεργά στον προγραμματισμό αυτής της ενημερωτικής εκστρατείας για την καταπολέμηση της βίας στην οικογένεια στην Ευρωπαϊκή Ένωση, αξιοποιώντας τις καλές πρακτικές της Πολωνίας, μεταξύ άλλων και την ε, δική μας εκστρατεία «Αγαπώ, δεν χτυπώ». Η ενημερωτική εκστρατεία θα ξεκινήσει φέτος το Σεπτέμβριο στην Πολωνία με διάφορα τηλεοπτικά σποτ, στα οποία συμμετέχουν διεθνείς κινηματογραφικοί αστέρες και κατόπιν καταιγιστικά θα συνεχιστεί αυτή η εκστρατεία στις χώρες μέλη που έχουν δηλώσει συμμετοχή. Και μάλιστα η εκδήλωση που θα ολοκληρώσει την ευρωπαϊκή αυτή εκστρατεία θα είναι μια διεθνής διάσκεψη που θα οργανωθεί στην Πολωνία τον Δεκέμβριο του 2011. Σε ό,τι αφορά τώρα τις ε, νομοθετικές ε, προτάσεις, η Πολωνία θα συνεχίσει τις εργασίες της για την αναθεώρηση της οδηγίας για τη μητρότητα, όπως αναφέρεται. Θα εξετάσουμε περαιτέρω τρόπους ε, και ρυθμίσεις λαμβάνοντας υπόψη ότι για πολλά χρόνια οι υποχρεώσει αυτής της οδηγίας οδήγησαν τα κράτη-μέλη σε υιοθέτηση νομικών διατάξεων προκειμένου να εξασφαλίσουν τις προδιαγραφές και τις απαιτήσει οδηγίας, αλλά ο τρόπος με τον οποίο επέλεξαν να συμμορφωθούν με την οδηγία είναι πολύ διαφορετικός. Έτσι εξηγούνται οι διαφορές που υπάρχουν στις εθνικές νομοθετικές διατάξεις για το θέμα αυτό. Δεν μας εκπλήσει αυτή η διαφορά γιατί κάθε χώρα επέλεξε διαφορετικό τρόπο για να συμμορφωθεί με την οδηγία αυτή για τη, για τη μητρότητα. Έχουμε την αίσθηση ότι αν θέλουμε να έχουμε την ευκαιρία να καταλήξουμε στη συμβαστική λύση, θα πρέπει να προτείνουμε κάποια μέτρη, κάποιες ρυθμίσεις που θα σέβεται στο μέτρο του δυνατού αυτή την ποικιλομορφία των μοντέλων της προστασίας των δικαιωμάτων της μητρότητας στα κράτη-μέλη και γενικώ των δικαιωμάτων ε, των γονιών. Από αυτή την άποψη η Πολωνία ε, πρόκειται να προσκαλέσει τους υπουργούς σε μια άτυπη ανταλλαγή απόψεων, εμπειριών και καλών πρακτικών στη διάρκεια του άτυπου Συμβουλίου Υπουργών. Μάλιστα ε, ευελπιστούμε ότι η συζήτηση αυτή θα επιτρέψει ένα νέο άνοιγμα στις εργασίες για την οδηγία αυτή. Θα ήθελα και πάλι να σας ευχαριστήσω θερμά για την προσοχή και σας προσκαλώ στις οργανώσεις και στις εκδηλώσεις ε, της Πολωνικής Προεδρίας, σε αυτές που θα γίνουν στην Πολωνία και στην διάσκεψη των εμπειρογνωμόνων και στις διάφορες άλλες οργανώσεις και εκδηλώσεις που θα γίνουν για την προώθηση της ισότητας των δύο φύλων και σε θέματα απασχόλησης αλλά και σε θέματα κοινωνικής πολιτικής. Σας ευχαριστώ. Eh, ευχαριστώ κυρία ε, Υπουργέ για την πληροφόρηση. Σας ευχαριστώ συγχρόνως και για την ε, πρόσκληση την οποία απευθύνατε σε όλους. Και τώρα θα ήθελα να καλέσω την κυρία Ελσβιέτα Ρατζιτζεύκα να λάβει τον λόγο. Είναι η πληρεξούσιος της πολιτικής κυβέρνησης για την ίση μεταχείριση. Σας ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Καλησπέρα σας. Και σας ευχαριστώ θερμά για αυτή την πρόσκληση στην σημερινή συνεδρίαση της Επιτροπής Δικαιωμάτων της Γυναίκας. Πιστεύω ότι εγώ ως πληρεξούσιος της πολωνικής κυβέρνησης για την ίση μεταχείριση οι εργασίες και προσπάθειες του, του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου για το θέμα αυτό είναι πολύ σημαντικέ και ε, τυχάνουν ιδιαίτερη προσοχή οι προσπάθειε σα και οι προτάσεις και στην Πολωνία. Όπως μας είπε και ο Υπουργός Φέντακ, στη διάρκεια της Πολωνικής Προεδρίας ε, θα γίνουν πολλές προσπάθειες για την καταπολέμηση της διακριτικής μεταχείρισης και θα ήθελα να αφαιρθώ στα θέματα της δικής μου αρμοδιότητας γιατί κάθε χώρα ε, αντιμετωπίζει με διαφορετικό τρόπο αυτή την προσπάθεια αποκατάστασης της ισότητας. Στην Πολωνία, ο θεσμό του πληρεξούσε τη πολωνική κυβέρνηση ε, ξεκίνησε το Μάρτιο του 2008 και ήταν ε, ε, άνευ προηγουμένω στην πολωνική ιστορία. Πρώτη φορά προβλέψαμε αυτό το πληρεξούσιο. Προηγουμένω είχαμε πληρεξούσιο για τι γυναίκε και τα παιδιά, τι γυναίκε και την οικογένεια. Και μάλιστα για τέσσερα χρόνια είχαμε πληρεξούσιο τη κυβέρνηση για την ίση κατάσταση ανδρών και γυναικών. Αλλά δεν είχαμε ποτέ πληρεξούσιο τη πολωνική κυβέρνηση για την ίση μεταχείριση. Ο Πρωθυπουργός μας όμως ήθελε το θέμα της μεταχείρισης να το θέσει ως οριζόντιο ζήτημα όλων των Υπουργείων και της κυβέρνησης. Γι' αυτό και ο πληρεξούσιος ε, της πολωνικής κυβέρνησης ακριβώς υπάγεται, βρίσκεται υπό την αιγίδα του ίδιου του, ίδιου του Πρωθυπουργού και φυσικά το έργο λαμβάνεται υπόψη και στα 17, προεδρία, στα 17 συγγνώμη, Υπουργεία και μας ενδιαφέρει στενή συνεργασία, παρακολούθηση των διαφόρων κυβερνητικών πράξεων και οι συγκεκριμένες δραστηριότητες και συνεργασίες με τα μεμονωμένα Υπουργεία και όπου απαιτείται διυπουργική συνεργασία έχουμε και μια διυπουργική μονάδα που απαρτίζεται είτε από τρει, τέσσερι, εφτά υπουργού, ανάλογα με το πρόβλημα, με τη φύση του προβλήματο και τα υπουργεία που εμπλέκονται. Και μάλιστα εγώ κάνω μια υποπτία και έχω και κάποιε δραστηριότητε συντονισμού και συνεργασία και προσωπικά με τα διάφορα υπουργεία. Από την 1η Πρώτου του 2011 τέθηκε σε ισχύ ο νόμο για την εφαρμογή τη Οδηγία Ευρωπαϊκή Ένωση ε, με βάση την, το νομικό καθεστώς του πληρεξούσιου τη πολωνική κυβέρνηση. Γιατί το, το 2008 είχαμε ε, κανονισμό του Συμβουλίου Υπουργών, τώρα έχουμε ειδικέ αρμοδιότητες του πληρεξούσιου τη πολωνική κυβέρνηση και μάλιστα δικαιούται να προτείνει και νομοθετικέ ε, πράξει. Δηλαδή συμμετέχει κατά κάποιο τρόπο στην νομοπαρασκευαστική προσπάθεια τη κυβέρνηση. Και μάλιστα ο πληρεξούσιο τη κυβέρνηση, στα πλαίσια τη συνεργασία, μπορεί να συγκροτήσει ομάδε εμπειρογνωμόνων με συμμετοχή ε, μη κυβερνητικών οργανώσεων ε, από διάφορα υπουργεία και επίση μπορεί να συγκροτήσει κάποιε μεικτέ ομάδε που θα παρτίζονται από εκπροσώπου τη κυβέρνηση, τη αυτοδιοίκηση, δηλαδή κρατικών και περιφερειακών αρχών, από εκπροσώπους μη κυβερνητικών οργανώσεων, από διάφορα Ινστιτούτα και φορείς, αλλά να προσκαλέσει και ανεξάρτητους εμπειρογνώμονες. Και τέτοιου είδους ε, ομάδες υπάρχουν πολλές. Θα σας ε, αναφέρω τώρα τρία πιο σημαντικά πράγματα, πιο σημαντικές προτεραιότητες της Πολωνικής Προεδρίας. Ε, θα είμαστε μια φθινοπορεινή Προεδρία, γι' αυτό και θα οργανώσουμε την πέμπτη Σύνοδο Κορυφής της Ισότητας που θα γίνει στο Πόσναν τον Νοέμβριο του 2011 και επειδή εγώ ασχολούμαι με την καταπολέμηση της διακριτικής μεταχείρισης σε όλα τα μέτωπα. Θέλουμε πραγματικά να εφαρμόσουμε αποτελεσματικά την αρχή της ίσης μεταχείρισης και στα πλαίσια καλών πρακτικών και ανταλλαγής απόψεων προκειμένου να έχουμε αποτελεσματική εφαρμογή της ίσης μεταχείρισης και στο δημόσιο και στον ιδιωτικό βίο, εμπλέκουμε όχι μόνο το επίπεδο το εθνικό, αλλά θέλουμε να φτάσουμε και πιο κοντά στον πολίτη, στο τοπικό και περιφερειακό επίπεδο. Γιατί περισσότερο ε, οι πολιτικέ σε περιφερειακό επίπεδο έρχονται κοντά στην πραγματικότητα των πολιτών. Γι' αυτό μας ενδιαφέρει η ανάμειξη όλων των επιπέδων και η συμμετοχή της αυτοδιοίκηση. Γιατί η αυτοδιοίκηση βρίσκεται κοντά στου πολίτε. Στην περίπτωση τη Πολωνία έχουμε μια μεγάλη χώρα ε, και πολλές εθνότητες. Για παράδειγμα, έχουμε κοινότητα Ρωμά σε διάφορα τμήματα της Πολωνίας. Επίσης, έχουμε πιστούς διαφόρων εκκλησιών. Τρεις είναι ε, οι βασικές, η Ορθόδοξη Καθολική Εκκλησία και η Ευαγγελική Λουθερανική Εκκλησία. Δηλαδή, έχουμε ε, ανθρώπους από διάφορες ε, θρησκευτικές ε, πεπιθήσεις ε, και εθνοτικές παραδόσεις. Θέλουμε λοιπόν να δράσουμε και με παιδαγωγικό ρόλο, να καταρρύψουμε κάποια στερεότυπα που μπορούν να οδηγήσουν σε προκαταλήψεις και διακριτική μεταχείριση. Γι' αυτό και αυτή τη σύνοδο κορυφής για την ισότητα θέλουμε να αναμίξουμε ενεργά και τις τοπικές και περιφερειακές αρχές, αξιοποιώντας περισσότερο το δυναμικό και των μη κυβερνητικών οργανώσεων, κυρίως από μικρούς δήμους και κοινότητες. Θέλουμε να δραστηριοποιήσουμε και τα μέσα μαζικής ενημέρωσης, τα τοπικά και γενικώ να γίνει μια ευαισθητοποίηση του ζωντανού ιστού της ε, πολωνικής κοινωνίας όσο πιο κοντά γίνεται στον πολίτη. Και θέλουμε αυτό που έχουμε θεσπίσει στον νόμο να το ε, εφαρμόσουμε και στην πράξη. Έχουμε και μία πλατφόρμα για τους Ρωμά που θα διοργανωθεί στις Βρυξέλλες για τα προβλήματα των Ρωμά. Οι Ρωμά ε, σήμερα αντιμετωπίζουν πολλά προβλήματα στην Ευρώπη και το ζήτημα των Ρωμά μας απασχολεί όλους. Στην Πολωνία δεν έχουμε τόσο οξύ πρόβλημα γιατί είναι πολύ μικρό το ποσοστό ούτε ένα δεκατό, αλλά σίγουρα και οι Πολωνοί Ρωμά αντιμετωπίζουν τα προβλήματα των υπόλοιπων Ρωμά και φυσικά ε, αντιμετωπίζουν αυτό το πρόβλημα του κοινωνικού αποκλεισμού. Είχαμε και ένα, πλαίσιο, ένα πρόγραμμα πλαίσιο για την κοινωνική ένταξη των Ρωμά στην Ευρωπαϊκή Ένωση και μάλιστα και για τις ομάδες Ρωμά υπάρχει πολλές φορές διαφορετική μεταχείριση. Η πιο περιθωριοποιημένη ομάδα μεταξύ των Ρωμά είναι οι γυναίκες Ρωμά. Μάλιστα ε, θα έχουμε τον ε, Απρίλιο την ημέρα του Ρωμά με διάσκεψη, συμμετοχή γυναικών Ρωμά από όλα τα μέρη της Πολωνίας. Και πολλές φορές ε, διαπιστώνουμε ότι οι γυναίκες είναι τελείως περιθωριοποιημένες, δεν έχουν ε, φωνή και γι' αυτό οργανώσαμε αυτό το φόρουμ στη Βαρσοβία για να δώσουμε φωνή και στις γυναίκες των Ρωμά για να δούμε ποια είναι η δική τους άποψη για το τι συμβαίνει στη δική τους ε, κατάσταση στον 21ο αιώνα και στην πλατφόρμα που θα γίνει στις Βρυξέλλες ε, θέλουμε να δώσουμε ιδιαίτερη φωνή στην, στο γυναικείο στρώμα των Ρωμά γιατί αυτές είναι οι πλέον περιθωριοποιημένες. Άλλο σημαντικό σημείο του έργου μας είναι η προσπάθεια συνέχισης ε, της οδηγίας. Η Γαλλική Προεδρία ξεκίνησε το 2008 τις εργασίες για αυτή την οριζόντια οδηγία. Φυσικά υπάρχουν ακόμη προβλήματα και πολλά οφείλονται και στην ε, παγκόσμια και ευρωπαϊκή οικονομική κρίση. Αλλά νομίζω ότι είναι πολύ καλή αυτή η οδηγία και θα πρέπει να συνεχίσουμε τι προσπάθειε, γιατί περιλαμβάνει ζητήματα και πέραν τη απασχόληση και τη αγορά εργασία που προηγουμένω δεν λαμβάνονταν υπόψη. αφορά την συμμεταχείριση ε, για λόγους ε, θρησκευτικούς, ε, εθνοτικούς, ε, γενετήσιου προσανατολισμού κτλ. Και νομίζω ότι είναι πολύ σημαντικό νομοθέτημα σε ό,τι αφορά την καταπολέμηση της διαφοροποιημένης και διακριτικής μεταχείρισης. Η Πολωνική Προεδρία θα συνεχίσει τις εργασίες για την οδηγία ίσης μεταχείρισης Επίσης μας ενδιαφέρει ιδιαίτερη θέση των ηλικιωμένων, γιατί είναι οξύ το δημογραφικό πρόβλημα που αντιμετωπίζει η Ευρώπη, αλλά και η Πολωνία. Εγώ είμαι γιατρός στο επάγγελμα και γνωρίζω ότι αυτό το ζήτημα είναι εξαιρετικά επώδυνο και για την πολωνική και την ευρωπαϊκή κοινωνία. Και σήμερα οι, οι άνθρωποι ζουν περισσότερο, οι άνδρες ε, ε, ζουν περισσότερο και οι γυναίκες ακόμη περισσότερο και οι, πολλές φορές οι ηλικιωμένοι άνθρωποι είναι μόνοι τους, απομονωμένοι, έχουν πολύ μικρή σύνταξη, είναι αβοήθητοι, άποροι, μακριά από την οικογένειά τους, μερικές φορές και άρρωστοι. Η κατάστασή τους είναι πραγματικά δίνη και πιστεύω ότι οι διατάξεις, ιδιαίτερα για τους ηλικιωμένου είναι πολύ σημαντικές. Μην ξεχνάτε ότι το επόμενο έτος ε, ε, θα ανακηρυχθεί το Ευρωπαϊκό Έτος των Ηλικιωμένων. Οπότε η προβληματική των ηλικιωμένων θα πρέπει να μας απασχολήσει ιδιαίτερα. Επίσης, ε, στις 2 Αυγούστου έχουμε την ημέρα που αφιερώνεται στο ολοκαύτωμα των Ρωμά. Είναι η ημέρα που θυμόμαστε την ε, εξουδετέρωση των Ρωμά ε, στο στρατόπεδο του Auschwitz και θα έχουμε επευκαιρία αυτής της ε, επαιτίου για δεύτερη φορά και Ρωμά από διάφορα μέρη του κόσμου και νομίζω ότι αξίζει να θυμόμαστε αυτό το επώδυνο βέβαια κεφάλαιο της ευρωπαϊκής ιστορίας δεν θα πρέπει να πέσει στη λύθη. Πολλές ε, οργανώσεις όπως βλέπετε θα γίνουν στη διάρκεια της Πολωνικής Προεδρίας. Θα ήθελα να σας απευθύνω έκκληση για συνεργασία και κατά της Πολωνικής Προεδρίας κατά τη διάρκεια της αλλά και μετά. Είμαι στη διάθεσή σας για να απαντήσω σε ερωτήσεις και απορίες. Περίμενα με μεγάλη ανυπομονή σε αυτή τη συζήτηση, αλλά ως γυναίκα εργαζόμενη βουλευτής Έχω μεγάλες προσδοκίες από το νομοθετικό έργο και από το ρόλο το βουλευτικό και τον ε, ρόλο του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και θαυμάζω το έργο της Επιτροπής σας ειδικά. Έχω δύο παρακλήσεις. Αν θέλουμε πραγματικά να καταπολεμήσουμε τη βία εις βάρος των γυναικών και αυτή την επιθετικότητα ε, και την σεξουαλική εκμετάλλευση των γυναικών, αυτή την ε, αντιμετώπιση της γυναίκας ως αντικείμενο και ιδιαίτερα σεξουαλικό αντικείμενο. Αν θέλουμε να καταπολεμήσουμε ε, αυτή τη στάση, θα ήθελα να σας ε, ε, επιστήσω την προσοχή στο ψήφισμα του Κοινοβουλίου του 2008 που αφορά τις διαφημίσεις και την εικόνα που δίνουμε για τις γυναίκες στις διαφημίσεις και για την εικόνα των αλλών, αλλά περισσότερο διαφημίσεις γίνεται εκμετάλλευση των γυναικών. Εδώ και δύο χρόνια η, οργάνωση, η κυβέρνηση προσπαθεί, ακολουθώντας αυτό το ψήφισμα, να διοργανώσει ε, διαγωνισμό μεταξύ των διαφημιστών, μεταξύ των διαφημιστών που προτείνουν τα διαφημιστικά σπότ και των πελατών τους, των αγοραστών. Και μάλιστα θα έχουμε και φεστιβάλ της διαφήμισης και σε αυτό το φεστιβάλ διαφήμισης θα δώσουμε βραβείο σε μια διαφήμιση που πραγματικά θα καταρρύπτει τα στερεότυπα της διαφήμισης. Και ειδικό βραβείο θα δοθεί για όλη την ενημερωτική εκστρατεία, ε, για τη διαφήμιση που καταρρύπτει τα στερεότυπα. Και ελπίζω και τα υπόλοιπα ευρωπαϊκά κράτη να ασχοληθούν πολύ σοβαρά με το ψήφισμα αυτό και να φροντίσουν να εφαρμόσουν και στην πράξη αυτό το σημαντικό ψήφισμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. Επίσης, καλό θα ήταν να γίνουν κάποιες μελέτες στην Ευρώπη και συζήτηση για την σεξουαλική εκμετάλλευση των παιδιών στην Ευρώπη και ιδιαίτερα των νεαρών κοριτσιών. Είναι μια άλλη μάστιγα και αυτή και παρακαλώ να μην ξεφύγει της προσοχής σας το θέμα αυτό, γιατί έχουμε όλο και μεγαλύτερη σεξουαλική εγκληματικότητα και σεξουαλική εκμετάλλευση των γυναικών, των παιδιών και ιδιαίτερα των νεαρών κοριτσιών. Σας ευχαριστούμε κυρία Ρατζησεύσκα. Τώρα θα έχετε την ευκαιρία να κάνετε ερωτήσεις και απαντήσεις. Είμαι βέβαιη ότι γνωρίζετε πως όλα αυτά τα ζητήματα είναι πολύ σημαντικά. Έχω πολλούς ομιλητές στον καταλογό μου. Θα ξεκινήσουμε δίνοντας λόγο στους συντονιστές των διαφορών πολιτικών ομάδων. Έχουν τρία λεπτά οι μικρότερες ομάδες θα έχουν 2,5 λεπτά. Ξεκινάω λοιπόν δίνοντας το λόγο στην κυρία Μπάουερ. Έχει 3 λεπτά. Και κάνω έκκληση σε όλους τους συναδέλφους. Παρακαλώ τηρήστε τους χρόνους. ότι στη στρατηγική 2020 υπάρχουν, υπάρχει ο πολύ φιλόδοξος στόχος ε, αύξησης τη ηλικία απασχόλησης και από την άλλη πλευρά ε, γνωρίζουμε ότι οι γυναίκες άνω των 50 ε, έχουν μικρές πιθανότητες να βρουν νέα απασχόληση. Αναφέρατε επίσης το στόχο σας για να αντιμετωπίσετε αυτό το ζήτημα πέρα από τα σχόλιά σας ε, όσον αφορά την ε, εξέβρεση συμβιβαστικών λύσεων θα ήθελα να τονίσω ότι πέραν των διαφορετικών πρακτικών το κυριότερο ζήτημα είναι τα διαφορετικά συστήματα χρηματοδότησης των αδειών μητρότητας. Θα ήθελα λοιπόν να σας ρωτήσω ποια είναι η δική σας άποψη, πώς θα βρεθεί η συμβιβαστική λύση για αυτό το ζήτημα ένα άλλο μεγάλο ζήτημα είναι επίσης η άδεια πατρότητας. Δεν θέλω καν να ανοίξω άλλα ζητήματα, διότι φαντάζομαι ότι αυτά θα συζητηθούν και από τους συναδέλφους μου. Η τελευταία ερώτηση. Είμαι πολύ ευχαριστημένη που αποφασίσατε να ασχοληθείτε με ένα μηχανισμό καταπολέμησης ε, της διακριτικής μεταχείρισης. Θα ήθελα λοιπόν να σας ρωτήσω έχετε σκοπό να απευθυνθείτε σε διαφορετικούς ε, φορείς ε, που υπερασπίζονται την ίση μεταχείριση ή σκοπεύετε να απευθυνθείτε σε τοπικούς φορείς. Ένα άλλο ζήτημα ε, είναι η ισότητα των φύλων. Η... η διαφορά μισθών μεταξύ φύλων. Θα ήταν ενδιαφέρον να το εξετάσουμε 17 με 18 είναι οι συνεδρίες της Βρυξέλλες. Τέλος πάντων, έχω την αίσθηση ότι ε, ανοίγει πολλά πολλά σημαντικά ζητήματα. Ευχαριστώ κυρία Μπάουερ. Η επόμενη μιλήτρια είναι η κυρία Τόμσον. Έχετε τρία λεπτά. απ' όλα θα ήθελα να σας ευχαριστήσω πολύ για την πολύ ενδιαφέρουσα παρουσίασή σας. Ήταν πολύ όμορφη έκπληξη. Κοιτώντα το πρόγραμμα της Πολωνικής Προεδρίας δεν έβλεπα τίποτα για την ισότητα των φύλων και τώρα ανοίγεται ένα κουτί με πολλά σημαντικά ζητήματα. Θα ήθελα να σα ρωτήσω κάτι. Okay, εντάξει, κάνουμε συνεδριάσεις, μαθαίνουμε για όλα αυτά τα ε, σημαντικά ζητήματα. Ποιε είναι όμως οι φιλοδοξίε σας κατά τη διάρκεια της Προεδρίας σας. Τι νομοθεσία θα θέλατε να προάγετε ή να αποφασίσετε εδώ στα ε, ευρωπαϊκά όργανα. Μιλάτε για διαγενειακή αλληλεγγύη σαν ε, ως ένα πρωταρχικό ζήτημα για εσάς. Επίσης για την ε, βία και για την νομοθεσία κατά της βίας στην Πολωνία. Θα ήθελα λοιπόν να μου πείτε ποιες είναι οι δικές σας προοπτικές σε ευρωπαϊκό επίπεδο. Πότε μπορούμε να οριστικοποιήσουμε όλα αυτά. Και επίσης αναφέρατε την άδεια μητρότητας. Ε, έχουμε πολύ μεγάλες προσδοκίες από την Πολωνική Προεδρία. Μιλάτε για διαφορετικούς κανονισμούς όσον αφορά την άδεια μητρότητα στις διάφορες ευρωπαϊκές χώρες. Πιστεύω ότι ακόμη και στη δική μου χώρα, στη Δανία, η νομοθεσία είναι εξαιρετικά απερχαιωμένη. Τα δικαιώματα των γυναικών σε άδεια μετρότητας θεωρούνται ως πρόβλημα στην αγορά εργασίας που διαπραγματεύονται οι διάφοροι εταίροι της αγοράς εργασίας. Το δικαίωμα της άδειας μητρότητας έπρεπε να αποτελεί θεμελιώδες ανθρώπινο δικαίωμα στην νομοθεσία. Είναι σημαντικό να αλλάξουμε την νοοτροπία σε ορισμένα κράτη-μέλη. Επίσης, ε, ένα πολύ θετικό πράγμα που πιστεύω, όταν μιλήσετε για οριζόντια οδήγια, δεν έχουμε αποφασίσει ακόμα για την οδηγία σε σχέση με την οριζόντια οδηγία κατά των διακρίσεων, η οποία είναι απολύτως απαραίτητη. Μιλάτε ότι ορισμένε ομάδε ε, αντιμετωπίζουν περισσότερου αποκλεισμού από άλλου. Πώ ε, βλέπετε την κατάσταση των ομοφυλοφίλων στην Πολωνία και την ε, διακριτική του μεταχείριση. Επίσης, οι γυναίκες και τα αναπαραγωγικά δικαιώματα σε τρεις χώρες στην Ευρώπη οι γυναίκες δεν έχουν το δικαίωμα πρόσβασης σε εκτρώσεις. Σχεδιάζεται στην Πολωνία να διατηρήσετε τους αυστηρούς νόμους κατά των εκτρώσεων που ε, λόγω του οποίου οι γυναίκες πηγαίνουν, απευθύνονται στη Γερμανία και πολλές φορές δεν έχουν χρήματα για να πληρώσουν τις εκτρώσεις. Ευχαριστώ πολύ. Τώρα έχει το λόγο η κυρία Παβανόβα από την ομάδα ALDE. Πρόεδρε, ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστούμε τις Υπουργούς ε, για, για αυτή την πολύ ενδιαφέρουσα και μεγάλη παρουσίαση. Είναι εξαιρετικά φιλόδοξο σχέδιο για ένα εξάμεινο, αλλά ε, συνεργάζεται με τη Σουηδική και Ισπανική Προεδρία, συνεχίζεται με το ίδιο πνεύμα και ελπίζω ότι θα δώσετε ένα μεγάλο έργο ε, στη Δανέζικη Προεδρία. Έχω κάποιες ερωτήσεις ε, όσον αφορά κάτι που ανέφερε ήδη η κυρία Μπάουερ. Όσον αφορά την ε, ενεργό γύρανση, την παράταση του επαγγελματικού βίου, εδώ σε αυτή την Επιτροπή έχουμε συζητήσει ότι είναι αναγκαίο να υπάρχει μια ε, αντιμετώπιση προσανατολισμένη προς τα γέννη, προς τα φύλλα. Το υποστηρίζουμε κάτι τέτοιο και πιστεύουμε ότι θα ήταν μια καλή ιδέα να εξετάσουμε την ενεργογυρένση από άποψη φύλων ε, λαμβάνοντας υπόψη τα προβλήματα που αντιμετωπίζουν οι ηλικιωμένες γυναίκες όσον αυτό αφορά την ένδυα, το κοινωνικό αποκλεισμό. Όσον αφορά την άδεια θα ήθελα επίσης να μάθω κατά πόσο θα δεσμευτείτε. Δεν αποτελεί μυστικό ότι κατά τη Βελγική Προεδρία λόγω των βελγικών αρχών ε, είχαμε μία λίγο ε, μεροληπτική θέση και δεν μπορέσαμε να προχωρήσουμε ιδιαίτερα. Θα ήθελα να μάθω ποια θα είναι τα βήματα που θα λάβετε ενεργά ώστε να πείσετε τα υπόλοιπα κράτη-μέλη ότι θα πρέπει να εγκρίνουμε επιτυχώς αυτή την οδηγία. Η βία είναι επίσης ένα σημαντικό ζήτημα. Έχουμε δύο φακέλους σε αυτό το σύνολο κανόνα, αλλά όπως φαίνεται η Επιτροπή μας ε, έχει αποκλειστεί από το να συμπεριλάβει την ευκαιρία ε, από τα να συμπεριληφθεί σε ισότιμο επίπεδο. Θα θέλαμε να μας υποστηρίξετε δεδομένου ότι η Επιτροπή ΛΥΜΠΕ έχει ήδη αποφασίσει ότι δεν θα πρέπει να συνεργαστούμε οι Επιτροπές ΦΑΜ και ΛΥΜΠΕ αλλά ενδεχομένω θα μπορούσατε εσείς να αλλάξετε τη γνώμη σας ε, θετικά. Τέλος, ε, το gender mainstreaming είναι μια πρωτοβουλία που όπως φαίνεται έχει επιτυχία όταν μιλάμε όμως για γυναίκες στις επιχειρήσεις και στην πολιτική, η συμβολή των γυναικών στην οικονομική διακυβέρνηση θα πρέπει να ενισχυθεί. Σκοπεύετε να αναλύσετε περισσότερο αυτό το ζήτημα. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ κυρία Παβάνοβα. Ευχαριστώ κυρία Παβάνοβα και τώρα για δυόμιση λεφτά. Ευχαριστώ την κυρία ε, Φέντα και την κυρία Ρατζισεύσκα. Ε, πολύ με ενδιέφερε η παρουσίασή σας και χαίρομαι ότι παραμένετε εις ε, το θέμα της δραστήριας απασχολήσεως των γυναικών αλλά ότι τονίζετε ότι και οι γυναίκες που δεν εργάζονται πρέπει να θεωρηθούν και να αντιμετωπίζονται με τον ίδιο σεβασμό είναι ένα πρόβλημα το οποίο θα αντιμετωπίζουμε όλο και παραπάνω και είναι βασικό να επιτρέψουμε στις γυναίκες αυτές να γεράσουν με αξιοπρέπεια. Ένα από τα πιο βασικά θέματα ε, ήταν ε, ότι είπατε ότι σας αγαπώ άρα δεν σας χτυπήσω και είπατε ότι θα υπάρξει και ένα πρόγραμμα στην τηλεόραση με αστέρες ε, του κινηματογράφου. Θα ήθελα λοιπόν να τονίσω ότι αυτό είναι πάρα πολύ σοβαρό θέμα. Θα ήθελα να ξέρω τι κάνει η Πολωνία όσον αφορά τους πρόσφυγες, τα σχολεία για την ε, ε, ε, για τα παιδιά τον προσφύγων, για την αστυνομία, διότι δεν νομίζω ότι αυτό που μας χρειάζεται είναι ακριβώς η συμπαράσταση των αστέρων, και ένα άλλο θέμα είναι οι γυναίκες στον επαγγελματικό τομέα, σαν επιχειρηματίες. Είπατε ότι θέλετε να παραμένουν οι γυναίκες στις επιχειρήσεις. Τι κάνετε όμως για αυτές. Υπάρχει κάποια πρόβλεψη για μικροχρηματοδότηση, συνεχίζετε να τις βοηθάτε και τι κάνετε, ε, ε, ε, τι γίνεται στο θέμα της παιδείας. Επίσης, η συνάδελφος αναφέρθηκε στην γονική άδεια. Μπορείτε να μου πείτε τι συμβιβαστική λύση πιστεύετε ότι μπορείτε να επιτύχετε κατά την Προεδρία σας. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ κυρία Γιανακουδάκη. Και τώρα η κυρία Φιγκερέντο είναι η επόμενη. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Και εγώ θα ήθελα να αναφερθώ σε τρία-τέσσερα θέματα, εν συντομία, συνεχίζοντας τις σκέψεις και τις παρατηρήσεις και των προσκεκλημένων μας και των μελών της Επιτροπής μας. Θέμα πρώτο. Τα προβλήματα που αντιμετωπίζουν οι εργαζόμενες γυναίκες εν μέσω της κρίσης. Γιατί μέσα στην κρίση οι πρώτες που απολύονται, οι πρώτες που έχουν κακοπληρωμένες, επισφαλείς εργασίες ή που υφίστανται την ανεργία είναι οι γυναίκες. Είναι θύματα διακριτικής μεταχείρισης ε, ακόμη και εντός της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Έχουμε μια τεράστια διαφορά μισθών πολλές φορές ε, μεταξύ ανδρών και γυναικών για την ίδια εργασία. Ποια είναι η γνώμη σας γι' αυτό. Προτίθεστε να αναλάβετε κάποια πρωτοβουλία γιατί η φτώχεια που μαστίζει τις γυναίκες και τα παιδιά είναι μια πραγματικά θλιβερή πραγματικότητα που δυστυχώς αποκτά όλο και μεγαλύτερες διαστάσεις με τις πολιτικές της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Δεν μπορούμε να ξεχνούμε την σοβούσα κρίση και εγώ κατάγομαι από μια χώρα που υφίσταται τις πολιτικές των πακέτων διάσωσης, των πολιτικών λιτότητας, θα ήθελα λοιπόν να μου πείτε τη δική σας γνώμη για το θέμα αυτό. Η φτώχεια έχει επιδεινωθεί γιατί γίνεται μια επίθεση κατά των κοινοφελών υπηρεσιών, ιδιαίτερα στον τομέα της κοινωνικής ασφάλισης, της υγείας. Και αυτά τα προβλήματα δυστυχώς έχουν αντικτύπωση στην καθημερινότητα των γυναικών. Τι ιδέες έχει, τι πρωτοβουλίες πρόκειται να αναλάβει η Πολωνική Προεδρία για το θέμα αυτό. Και ένα άλλο πρόβλημα για την ε, σεξουαλική και αναπαραγωγική υγεία. Δυστυχώς ε, έχουμε ακόμη τέτοια προβλήματα σε πολλές χώρες, ακόμη και στην Πολωνία. Πώς λοιπόν αντιμετωπίζετε αυτή την κατάσταση, τι πρωτοβουλίες προτίθεστε να αναλάβετε, ώστε να ενισχυθούν τα δικαιώματα των γυναικών και να εξασφαλιστεί το δικαίωμα ελεύθερης επιλογής για τη ζωή και το σώμα τους, ιδιαίτερα στον τομέα της σεξουαλικής και αναπαραγωγικής υγείας. Ένα άλλο θέμα, συναφές με το προηγούμενο, αφορά την άδεια πατρότητες και μητρότητας. Μια και εξάντλησε σχεδόν το χρόνο μου, μία τελευταία ερώτηση. Θα λάβετε κάποια πρωτοβουλία κατά της βίας, συνεχίζοντας το έργο των προηγούμενων προεδριών για την προάσπιση των δικαιωμάτων των γυναικών. Ευχαριστώ κυρία Φιγκερέντο. Και ε, ευχαριστώ κυρία Φιγκερέντο. Τώρα λοιπόν προχωράμε εις ε, την ομάδα των ομιλητών όπου κάθε ομιλήτρια έχει χρόνο δύο λεπτών για να μπορέσουν να τεθούν όσο το δυνατόν περισσότερες ερωτήσεις και να έχουμε επαρκή χρόνο και για τις απαντήσεις. Καταρχήν η κυρία Εστρέλα για δύο λεπτά. Ευχαριστώ κυρία Πρόεδρε. Και εγώ θα ήθελα, όπως και οι σα να ευχαριστήσω τις Υπουργούς για την παρουσία τους και την περιστατωμένη και πλήρη παρουσίαση που μας έκαναν για τις πολωνικές προτεραιότητες. Η Υπουργός μας μίλησε για πολύ σημαντικά θέματα όπως ε, το δημογραφικό πρόβλημα, την ενδοοικογενειακή βία, το συνδυασμό του επαγγελματικού και του οικογενειακού βίου για τις γυναίκες και για τους άντρες. Πολύ σημαντικά όλα αυτά τα θέματα. Αλλά όπως είπαμε και χθε στην Επιτροπή Απασχόλησης και Κοινωνικών Υποθέσεων, θα ήθελα να επανέλθω σε ένα θέμα που μου είναι ιδιαίτερα προσφυλές και αφορά την άδεια μητρότητας. Γιατί είμαι εισηγήτρια αυτής της πολύ σημαντική έκθεσης για την άδεια μητρότητα. Όπως διαπιστώστε κι εσείς, είναι πολύ υψηλέ οι προσδοκίε τη επιτροπή μας από την Πολωνική Προεδρία και το έργο που ελπίζουμε ότι θα επιτελέσει υπέρ της οδηγίας αυτής. Μάλιστα είχα την ευκαιρία και προηγουμένως ε, να μιλήσω και με σας κύριε Υπουργέ και με τον Υφυπουργό Κοινωνικών Υποθέσεων και να σας πω ότι Έχω υψηλές προσδοκίες από την Πολωνική Προεδρία γιατί η Πολωνία πραγματικά νομοποιείται να έχει πιο φιλόδοξες απαιτήσει από το Συμβούλιο, πολλά δε μάλλον που πρόσφατα αναθεώρησε την εθνική της νομοθεσία για το θέμα αυτό της άδεια μητρότητας και πατρότητας. Επίσης θα ήθελα να σας διαβεβαιώσω για την αμέριστη υποστήριξη του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και την προθυμία μας να συνεργαστούμε για να βρούμε κοινή λύση. Μάλιστα, πρόκειται να υποβάλουμε και προφορική ερώτηση με συζήτηση στο Συμβούλιο για να δώσουμε περισσότερο κουράγιο και δύναμη και στήριξη στην, Ευρωπαϊκή, στην Πολωνική Προεδρία για να πούμε ότι το θέμα δεν έχει κλείσει και ευελπιστούμε σε αίσια αποτελέσματα. Και ελπίζουμε στο άτυπο Συμβούλιο Υπουργών να επιτευχθεί συμφωνία, να βρεθεί η συνένεση για να έχουμε μια θετική εξέλιξη στο ζήτημα της άδειας μητρότητας. Ευχαριστώ. Και τώρα η κυρία Ζηλεύσκα για δύο λεφτά. Ευχαριστώ και ευχαριστώ θερμά και την κυρία Υπουργό και την Πληρεξούσιο για τα πολύ αυτά σημαντικά θέματα και τις προτεραιότητες της Πολωνικής Προεδρίας. Θα ήθελα να σας διαβεβαιώσω, κυρία Στρέλα, ότι σίγουρα οι Πολωνοί Ευρωβουλευτές είναι ένθερμοι υπέρμαχοι της οδηγίας για την άδεια και μάλιστα εμείς στην Πολωνία έχουμε πολύ πιο προηγμένες διατάξεις από ότι ορισμένες από τις διατάξεις της οδηγίας. Θα σας στηρίξουμε πλήρως και ευελπιστούμε ότι στη διάρκεια Πολωνικής Προεδρίας θα βρεθεί συμβαστική λύση για την οδηγία αυτή, ώστε να ε, γιορτάσουμε αυτή την ε, ευρωπαϊκή επιτυχία για την αποκατάσταση ίσων ε, δικαιωμάτων μεταξύ ανδρών και γυναικών. Η Φε, κύριε Υπουργέ, κυρία Φέντακ, η οδηγία αυτή αφορά την άδεια πατρότητα και άδεια μητρότητα. Αλλά εγώ θα ήθελα να σα μιλήσω για την άδεια υιοθεσία, γιατί ε, εγώ είμαι ε, υποστηρίκτρια των οικογενειών αυτών που δεν μπορούν να έχουν ε, δικά τους βιολογικά παιδιά και πριν από λίγα χρόνια βελτιώθηκε η σχετική πολωνική νομοθεσία για τις υιοθεσίε και σήμερα και όσοι υιοθετούν μπορούν να επωφεληθούν από την άδεια και μάλιστα η Πολωνική Προεδρία νομίζω ότι ετοιμάζει και νέα μέτρα. Καλό θα ήταν να εξομοιώσουμε αυτές τις άδειες για να έχουμε ίσα δικαιώματα σε όλα τα κράτη-μέλη. Κυρία Υπουργέ Φέντακ, με ποιο τρόπο πρόκειται η Πολωνική Προεδρία να ενισχύσει τη συμμετοχή των γυναικών στην αγορά εργασία. Γίνονται συζητήσει για τι ποσοστώσει, για την ενίσχυση στα διοικητικά συμβούλια των επιχειρήσεων κτλ. Θέλω τη θέση λοιπόν τη Προεδρία για το θέμα αυτό. Και τέλο, κυρία Υπουργέ Ραζισεύσκα, θα ήθελα να μιλήσω για την ε, διακριτική μεταχείριση των γυναικών στον αθλητισμό πολύ συχνά ε, οι αθλήτριες ε, αμείβονται πολύ χαμηλότερα από τους ε, άνδρες συναθλητές τους. Υπάρχουν κάποια σχέδια της Πολωνικής Προεδρίας για να καλυφθεί και αυτή η αδικία. Η κυρία Γκουρμάη. Ευχαριστώ πολύ. Μεγάλη μου ευχαρίστηση άκουσα και τις δύο σας πολύ προσεκτικά. Χαίρομαι που κατά την ε, τριπλή προεδρία ε, βρήκα συγκεκριμένα θέματα συμβιβασμό της ε, επαγγελματικής και ιδιωτικής ζωής στην Ε, Πιστεύω ότι πρέπει οπωσδήποτε να επικεντρωθούμε στο gender mainstreaming σε οποιονδήποτε από αυτούς τομείς. Όσον αφορά την εξάλληψη της ένδυας, θα ήθελα να μάθω αν η Πολωνική Προεδρία σκέφτεται ότι υπάρχει κάποιο κομμάτι του πληθυσμού στο οποίο υπάρχουν προβλήματα όσον αφορά τις συντάξεις και αν θεωρούν ότι υπάρχει, πρέπει να λυθούν μέτρα ειδικά για τις γυναίκες ή υπάρχει ακόμα υψηλό ποσοστό ένδυας ειδικότερα για τις γυναίκες θα ήθελα να μην υπάρχουν πια ε, σύντομα ε, φτωχές γυναίκες Όσον αφορά την οδηγία της ίσης μεταχείρισης, πώς η Προεδρία σας βλέπει αυτή την απόφαση, τι παρακολούθηση πιστεύετε ότι θα γίνει, θέλετε να τροποποιηθεί η οδηγία αυτή και όπως μόλις τελείωσε η Ουγγρική Προεδρία ως Ούγγρος πολίτης χαίρομαι που μιλάτε για ολοκληρωμένη Προεδρία Ελπίζω ότι με αυτή την έκφραση συμπεριλαμβάνεται και τις γυναίκες. Ο Σουγκαρέζα θέλω να σε ευχηθώ καλή επιτυχία. Έχετε μεγάλες φιλοδοξίες και μπορείτε να υποστηρίζετε στην υποστήριξη του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. Ευχαριστώ πολύ για την πρόσκλησή σας και ελπίζουμε ότι η Πολωνική Προεδρία θα είναι φιλική προς το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και προς τις γυναίκες. Ευχαριστώ πολύ κύριε Γκούντουε. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ κυρία Μπόσχουτ, ευχαριστώ κυρία Πρόεδρε, ευχαριστώ για την εισαγωγή σας και ουσιαστικά έχω τρεις ερωτήσεις. Η πρώτη ερώτηση είναι για την ε, οδηγία κατά των διακρίσεων, μια οριζόντια ερώτηση, μετά ε, το θέμα της εξέτασης στο Κοινοβούλιο και εφόσον πρόκειται για άτομα τα οποία ζουν στην Πολωνία, για ε, ηλικιωμένοι νέοι, διακρίσεις βάσει του φύλου ή της και της ομοφιλίας. Ποια θα είναι η θέση σας κατά την Προεδρία για να δείξετε ότι ε, θέλετε να λύσετε τα θέματα αυτά. Επίσης το πακέτο των θυμάτων διότι αυτό που θα ήθελα να σας ρωτήσω είναι ε, ε, αν αναφέρεστε και στην, ε, στον ακροτηριασμό των γεννητικών οργάνων των γυναικών διότι είναι θέματα τα οποία απασχολούν όλη την Ευρωπαϊκή Ένωση και χρειάζεται μια ευρωπαϊκή πολιτική επ' αυτού. Η τρίτη ερώτηση αναφέρεται σε την πρόσβαση σε θέσεις υψηλού επίπεδου και συμφωνώ και εγώ ότι είναι κάτι πολύ βασικό και εφόσον η Πολωνία θα οργανώσει το 2012 το Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα Ποδοσφαίρου θέλω να ρωτήσω για τα αθλητικά. Ξέρετε ότι σε, ορισμένα, σε ορισμένους οργανισμούς δεν υπάρχει σχεδόν καμία γυναίκα ε, γιατί θέλω να επιστήσω την προσοχή σας και νομίζω ότι είναι κατάλληλη στιγμή να το συζητήσετε και να το επιδιώξετε. Και τέλος, στο Συμβούλιο ε, θα υπάρξει ένα εργαστήριο για το πώς φίλοι υπάρχουν. Θα συζητήσετε και τα προβλήματα ε, των των ε, ενδιαμέσων φίλων κατά αυτή τη διάρκεια. Η κυρία Παπαδοπούλου τελευταία. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ. Ε, θέλω να ευχαριστήσω τις τρεις προεδρίες, ε, την ε, Πολωνία την, και την Κύπρο που είναι η δικιά μου χώρα και θεώρησα ότι η ισότητα των φύρων είναι δικό σας θέμα. Θα ήθελα πιο συγκεκριμένα ε, βήματα όμως και αυτή είναι η πρώτη μου ερώτηση. Η δεύτερη ερώτηση αναφέρεται στις διεθνείς συμφωνίες διότι από ό,τι γνωρίζω η Πολωνία έχει δεχθεί χωρίς επιφυλάξεις διάφορες ε, διεθνείς συμφωνίες ε, του Πεκίνου, του Καΐρου γιατί η Πολωνία δεν εφαρμόζει αυτές τις αποφάσεις όπως έχουν συστήσει διαφορεί και τρίτον το ερώτημα είναι σχετικά με τη στρατηγική της κυβερνήσεως. Στην Πολωνία υπάρχει μία κυβερνητική πολιτική για την ισότητα των φύλων και αν όχι πότε πρόκειται να συμβεί αυτό. Ευχαριστώ πολύ. Και τώρα κυρία Χιμένας. Ευχαριστώ. Και ευχαριστώ και τις εκπροσώπους τη Πολωνική Προεδρίας ε, για τις εξαιρετικέ ε, παρουσιάσεις που μας έκαναν, για τις προκλήσεις τη πολωνική Προεδρίας στο επόμενο εξάμεινο. Αναφερθήκατε σε όλα τα θέματα που μας απασχολούν, που μας ενδιαφέρουν ε, και συνεχώς τα έχουμε στην ημερήσια διάταξη. Μεταξύ άλλων αναφερθήκατε και στην βία κατά των γυναικών. Ερωτώ για το θέμα της καταπολέμησης της βίας. Ποιες θα είναι οι πρωτοβουλίες της Πολωνικής Προεδρίας ό,τι αφορά την προώθηση ε, της Ευρωπαϊκής Εντολής για την προστασία των θυμάτων. Γιατί ασχολήθηκα με την έκθεση αυτή που εγκρίθηκε το προηγούμενο Δεκέμβριο στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Κατόπιν η κατάσταση έφτασε σε αδιέξοδο. Τελικά ε, έχουμε λάβει την εντολή για να προχωρήσουμε στη δεύτερη ανάγνωση. Ερωτώ λοιπόν πώς έχουν τα πράγματα το στο Συμβούλιο. Θα ξεκινήσει ο τριμερής διάλογος, ποιο είναι το πρόγραμμα της Πολωνικής Προεδρίας ό,τι αφορά τι εργασίε για την Ευρωπαϊκή Εντολή Προστασία των Θυμάτων. Ευχαριστούμε κυρία Χιμένες. Κυρία Νέλα Ευχαριστώ κυρία ε, Υπουργέ. Ε, ξέρω ότι έχετε μεγάλες φιλοδοξίες, πολλά προγράμματα και ελπίζω θα μπορέσετε να επιτύχετε τουλάχιστον τα περισσότερα από αυτά. Έχω μία ερώτηση που αναφέρεται στην ισότητα των φίλων μεταξύ, με, στο, ισότητα των δικαιωμάτων μεταξύ των φίλων, ιδίω στο μισθό. Ε, και θα ήθελα να ξέρω τι συγκεκριμένα πρόκειται να κάνετε πέραν των σεμιναρίων θα ήθελα να γνωρίζω αν υπάρχει κάτι το οποίο προτίθεστε να κάνετε επί του θέματος και μετά η αναπαραγωγική υγεία και ο οικογενειακός προγραμματισμός. Μιλήσατε για τη σεξουαλικότητα των γυναικών, αλλά αν θεωρούμε ότι υπάρχει πρόβλημα πρέπει να μπορεί κανείς να το συζητήσει και εάν απαγορεύονται ακόμη οι αμβλώσεις στη χώρα σας πρέπει να σκεφτείτε τι βήματα θα έπρεπε να αναλυφθούν αυτό το οποίο δεν έχετε αναφέρει και μία ε, ε, συμβουλή ε, για τα σχολεία πρέπει ήδη στα μικρά παιδιά να εξηγεί κανείς τι είναι σωστό και τι είναι όχι πως μπορεί να προστατευτεί κανείς από μία κατά λάθο εγκυμοσύνη και εντός ορισμένων μηνών θα ήθελα να ξέρω ακριβώς τι επιτύχατε Ευχαριστώ Και τώρα η κυρία Πικβίτσα. Ευχαριστώ κυρία Πρόεδρε, ευχαριστώ και, τους δι... και τις δύο υπουργούς για την παρουσίασή τους και την παρουσίαση των προτεραιοτήτων για το ερχόμενο εξάμενο. Χαίρομαι ιδιαίτερα που βρίσκομαι εδώ και που μαθαίνω ότι η Πολωνία θα προβεί σε συγκεκριμένα βήματα για το ζήτημα της ισότητας των φύλων. Διαβάζοντας το πρόγραμμα της Προεδρίας δεν είδα κάτι τέτοιο και είχα στεναχωρηθεί. Ε, θα, θέλω, χαίρομαι που θα έχουμε την ευκαιρία να συνεργαστούμε και τους εύχομαι καλή τύχη στην επιτευξή αυτών των στόχων. Θέλω να ρωτήσω την Υπουργό, έχετε συγκεκριμένα σχέδια για το πώς θα επιτύχετε την ισότητα απόψη συντάξεων μεταξύ ανδρών και γυναικών. Αυτό αποτελεί σημαντικό ζήτημα για τις ηλικιωμένε γυναίκες όταν λαμβάνουν χαμηλότερες συντάξεις ε, πέφτουν στην παγίδα της ένδυας. Έχετε κάποια, προβλέψει κάποια συγκεκριμένα μέτρα. Δεύτερη ερώτηση. Χαίρομαι που η Πολωνία προσέχει ιδιαίτερα την εναρμόνιση της ιδιωτικής και επαγγελματικής ζωής της ιδιωτικής ζωής και της σταδιοδρομίας. Τι θα κάνετε για να βοηθήσετε τις γυναίκες να εργάζονται και ταυτόχρονα να έχουν μια ικανοποιητική ιδιωτική ζωή. Τρίτο ερώτημα. Πρέπει να βρούμε μέτρα για να καταπολεμήσουμε την παιδική ένδικη. Το επίπεδο αυτής αυξάνεται διαρκώς και δεν έχουμε καταφέρει να το μειώσουμε. Τέλος, ε, θα ήθελα να ευχηθώ καλή τύχη στην Πολωνία. Αν καταφέρει να ολοκληρώσει τις εργασίες ε, για αυτή την οδηγία και να αντιμετωπίσει ε, τα ζητήματα ε, της ισότητας των φύλων. Ευχαριστώ πολύ. Η επόμενη μιλήτρια, κυρία Ζαμπόρσκα. Ευχαριστώ κυρία Πρόεδρε. Ευχαριστώ για την εισαγωγή που κάνατε ε, και οι δύο εκπρόσωποι της Πολωνίας και θέλω να ε, αντιδράσω αυτά που είπε η κυρία Παπαδοπούλου που είπατε ότι σχετικά με τις γυναίκες πρέπει να τους διευκολύνεται την πρόσβαση στην αγορά εργασίας ιδίως στις πλέον ηλικιωμένες. Ε, κατά την περίοδο της οικονομικής κρίσεως υπάρχουν όλο και περισσότεροι άνεργοι και σε μια ε, πολύ άσχημη κατάσταση είναι ιδίω οι γυναίκες οι οποίες είναι κοντά στην ε, ηλικία συνταξιοδοτήσεως και έχασαν την εργασία τους. Είπατε ότι οι γυναίκες χρειάζονται μια αλληλεγγύη μεταξύ των γενιών και πιστεύω ότι υπάρχει και μια πολύ μεγάλη ομάδα γυναικών οι οποίες πριν τις συνταξιοδότηση ε, είναι ε, ήδη ε, πρέπει ακόμη να φροντίζουν τους γονείς τους και ίσως και τους, τη δεύτερη γενιά. Οπότε θα ήθελα να ξέρω αν θα μπορούσε να γνωρίσει κανείς επισήμως ότι η παρακολούθηση και περίθαλψη των μελών της οικογένειας ε, είναι ε, μια εργασία η οποία πρέπει να αμείβεται ικανοποιητικά, να καλύπτεται από την κοινωνική ασφάλιση ε, και να συνυπολογίζεται για την σύνταξη, πράγμα από το οποίο θα μπορούσε να βοηθήσει πολλές γυναίκες και να βελτιώσει την ε, θέση τους διότι πολλές φορές ε, είναι άνεργες και πρέπει ε, επίσης να μην απομονωθούν. Ευχαριστώ. Προτού δώσω το λόγο τώρα στις δύο μιλήτριες για να απαντήσουν θα ήθελα να ρωτήσω αν υπάρχει κάποιος άλλος που θέλει ακόμη να υποβάλει μία ερώτηση. Αν όχι θα ήθελα να στραφώ προς τις δύο φιλοξενούμενους μου και καταρχήν να δώσω το λόγο στην ε, κυρία Φέντα, η οποία έχει 8 λεπτά στη διάθεσή της για να απαντήσει σε όλα τα ερωτήματα που της τέθηκαν. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ, ευχαριστώ όλους όσους έθεσαν τις ερωτήσεις. Τι να προλάβει κανείς να απαντήσει μέσα σε 8 λεπτά πώς θα απαντήσει σε μια πληθώρα ερωτήσεων. Θα προσπαθήσω να ομοδοποιήσω τις ερωτήσεις, γιατί όντως σε μερικές ε, περιπτώσεις ε, οι ερωτήσεις αφορούσαν το ίδιο ζήτημα και υπήρχε μια αλληλοσυμπλήρωση. Πολλές ερωτήσεις τέθηκαν για την οδηγία για την άδεια μητρότητας. Είναι μια από τις ε, οδηγίες που βρίσκονται στο επίκεντρο του ενδιαφέροντος των εργασιών της Επιτροπής σας. Και η κυρία Εστρέλα, αλλά και άλλες ε, συνάδελφοι μίλησαν για το θέμα αυτό της οδηγίας και πόσο προσφυλής ε, τους είναι η προοπτική της προόδου στις εργασίες αυτής της οδηγίας στη διάρκεια της Πολωνικής Προεδρίας. Ας μην ξεχνούμε ότι στην Πολωνία σημειώσαμε αισθητή πρόοδο για τα θέματα άδεια μητρότητα. Στην αρχή της κοινοβουλευτική μα θητεία παρατείναμε ε, σημαντικά την ε, άδεια μητρότητα και μάλιστα παρατείναμε και την άδεια πατρότητα. Οπότε αυτή την άποψη πολλά άλλαξαν προς την καλή κατεύθυνση στην Πολωνία. Βέβαια, έχουμε ε, συνείδηση και επίγνωση τη δυσκολία αυτών των εργασιών. Δεν θα είναι καθόλου εύκολο για την Πολωνική Προεδρία να προωθήσει αυτό το θέμα. Πάντως είναι ε, έτοιμη και πρόθυμη να μην φυστεί προσπαθειών για να προωθήσει τι εργασίε και στη συνεργασία με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και το Κοινοβούλιο για την οδηγία αυτή. Βέβαια, έχουμε επίγνωση του γεγονότος ότι το βάρος του ζητήματος αυτού για την κοινωνική πολιτική της Ευρωπαϊκής Ένωσης είναι πολύ μεγάλο. Συνεχίζουμε τις διαβουλέψεις. Οι διαβουλέψεις ε, θα καλύψουν ε, την οδηγία και θα συμμετέχουν σε αυτές το Κοινοβούλιο, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ή οι ενδιαφερόμενες πλευρές. Θα γίνουν ευρύτατες διαβουλεύσεις για την οδηγία αυτή. Και Στόχος μας είναι να βρούμε έναν τρόπο να σημειώσουμε πρόοδο σε αυτό το κρίσιμο ζήτημα. Θα ήθελα πάντως να υπογραμμίσω ότι υπάρχουν μεγάλες διαφορές μεταξύ των εθνικών συστημάτων και πολλές αλλαγές έχουν γίνει στα εθνικά συστήματα, αλλά σίγουρα αυτές οι διαφορές θα έχουν κάποια επιρροή στην πρόοδο των εργασιών πετένα ένα άτυπο Υπουργικό Συμβούλιο το φθινόπωρο, 20 ε, και 21 Οκτωβρίου στην Κρακοβία και εκεί θα προσπαθήσουμε να προωθήσουμε αυτές τις ε, διαβουλεύσεις, την ανοιχτή συζήτηση και την ε, ανταλλαγή απόψεων και πρακτικών. Ελπίζω εκεί πραγματικά να γίνει κάποια πρόοδος ως προς την οδηγία. Έχουμε προβλέψει και συσκέψεις εργασίας για να εξοικειωθούμε με τις θέσεις των διαφόρων πλευρών, αλλά γνωρίζουμε ότι οι διαφορές δεν είναι μόνο διαδικαστικές ή οργανωτικές. Δυστυχώς είναι και ουσιαστικές διαφορές εξαιτία της δινής οικονομικής και δημοσιονομικής κατάστασης που αντιμετωπίζουν τα κράτη-μέλη. Και ίσως μπορέσουμε να βρούμε κάποια λύση στην οδηγία αυτή, προτείνοντας κάποια μέτρα, κάποιες διατάξεις που επίσης θα είναι ελαστικά και που θα σέβονται όσο περισσότερο γίνεται τα διάφορα ε, και τα πολύ περίπλοκα και πολύμορφα μοντέλα της προστασίας των δικαιωμάτων της μητρότητας που εφαρμόζονται στα διάφορα κράτη. Ίσως εκεί δεν βρεθεί η λύση από ένα σεβασμό των εθνικών διαφορών. Πάντως, η πρόοδος θα εξαρτηθεί από το πόσο διαλλακτική και συνεργάσιμη θα είναι στη συζήτηση οι συμμετέχοντες. Τώρα, σε ό,τι αφορά την ρήτρα, την ειδική ρήτρα και την ελαστικότητα, πιστεύω ότι θα μας υποστηρίξει το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Τώρα, για την άδεια πατρότητας, ή μάλλον για την άδεια υιοθεσίας, Η κυρία Σξιδλεύσκα, Υπέβαλε τη σχετική ερώτηση. Αναφυσβήτητα, η ρύθμιση θα πρέπει να είναι ίδια και για την άδεια μητρότητας και για την άδεια πατρότητας και για την άδεια υιοθεσίας. Θα πρέπει να γίνει μια εξομοίωση των δύο ή τριών αδειών. Άδειες μητρότητας κυρίως και άδεια υιοθεσίας όπως έγινε και στην Πολωνία. Τώρα, σε ό,τι αφορά το αδιέξοδο ή την πρόοδος προς την οδηγία, αυτό που είναι ε, σημαντικό είναι ότι σίγουρα ε, η πρόοδος είναι σημαντική, αλλά περισσότερο χρειαζόμαστε μια αλλαγή νοοτροπίας και μια προετοιμασία των, των κρατών μελών ώστε να δεχτούν τις νέες διατάξεις. Σε ό,τι αφορά την καταπολέμηση της ενδοοικογενειακής ε, βίας, εμείς επικεντρωνόμαστε στην προώθηση κάποιων ε, καλών διατάξεων και προώθηση καλών πρακτικών με ενημερωτικές εκστρατείες, με την καμπάνια αυτή που σας ανέφερα, προκειμένου να αλλάξει η νοοτροπία, να γίνει ένα είδος διαπαιδαγώγησης και αυτό το θέμα είναι πολύ σημαντικό με τη διαπαιδαγώγηση, την αλλαγή της νοοτροπίας μπορούμε να καταπολεμήσουμε αποτελεσματικά τη βία στο σπίτι. Τώρα, σε ό,τι αφορά το πακέτο για τη συμμετοχή, την ενίσχυση της συμμετοχής των γυναικών στην αγορά εργασίας, θα ασχοληθούμε και με τα τυπικά νομοθετικά σημεία και θα επιδιώξουμε συμπεράσματα σχετικά στο Συμβούλιο σε ό,τι αφορά το συνδυασμό του επαγγελματικού και του οικογενειακού βίου ανδρών και γυναικών. Προτεραιότητα της Πολωνίας είναι να διευκολύνει τους εργαζόμενους, άνδρες και γυναίκες, για να συνδυάσουν την επαγγελματική και οικογενειακή ιδιωτική του ζωή, ε, προβλέποντας μια ελαστικότητα στις διάφορες μορφές φροντίδας φύλαξη των παιδιών και διευκολύνοντας τη ζωή των εργαζομένων. Έχουμε καλή πείρα σε ό,τι αφορά την επιχειρηματικότητα των γυναικών, γιατί και αυτό αναφέρθηκε. Την τελευταία τετραετία υλοποίησαμε πολλά σχέδια ε, με θέμα την επιχειρηματικότητα των γυναικών, την ε, ίδρυση, την, ε, το άνοιγμα επιχειρήσεων εκ μέρους των γυναικών, την επαγγελματική δραστηριοποίηση των γυναικών και επίσης και στη διάρκεια της Πολωνικής Προεδρίας θα προωθήσουμε αυτά τα θέματα. Τώρα μιλήσατε για τη διάκριση βάρος των ηλικιωμένων. Το θέμα των ηλικιωμένων επίσης είναι προτεραιότητα της Προεδρίας μας. Αυτό σημαίνει ότι θα πρέπει να φροντίσουμε να εξασφαλίσουμε τις γυναίκες ε, και στην σύνταξη και μετά την ε, σύνταξη, γιατί εκεί σε εκείνη την φάση είναι πιο ευάλωτες στη φτώχεια. Και μάλιστα περιμένουμε εντός ολίγου την πράσινη βίβλο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για το θέμα των συντάξεων και θα συμμετέχουμε ενεργά στις συζητήσεις ε, για την πράσινη βίβλο γιατί σίγουρα το θέμα των συντάξεων και ιδιαίτερα των συντάξεων των γυναικών είναι πολύ σημαντικό. Το θέμα της ε, αμοιβή για την, για, για, την εργασία στο σπίτι επίσης είναι πολύ σημαντικό. Έχουμε αντίστοιχε ρυθμίσει και μέτρα και στην Εθνική Νομοθεσία. Και αν η Ευρωπαϊκή Επιτροπή τον Νοέμβριο ή και νωρίτερα τον Οκτώβριο, όπω ε, έχει αναγγείλει, υποβάλει την πράσινη βίβλο, Εμεί αμέσω θα ξεκινήσουμε τις εργασίε για το θέμα αυτό άλλη ερώτηση πώς ε, θα υλοποιήσουμε τους στόχους ε, ή πώς θα προωθήσουμε την υλοποίηση των στόχων της στρατηγικής του 2020 σε ό,τι αφορά την απασχόληση, την ισότητα σε θέματα απασχόλησης, ε, την καταπολέμηση της φτώχειας, πώς θα προωθήσει την υλοποίηση των στόχων η Ευρωπαϊκή Προεδρία. Σίγουρα θα συνεργαστούμε στενά με τα κοινοτικά θεσμικά όργανα και με τα κράτη-μέλη για να υλοποιήσουμε αυτούς τους στόχους, γιατί όλοι αυτοί οι στόχοι είναι θεμελιώδεις. Γι' αυτό και θα επιδιώξουμε την πραγματοποίησή τους. Θα προωθήσουμε και τις εμβληματικές πρωτοβουλίες. Για παράδειγμα, η Ευρωπαϊκή Πλατφόρμα Συνεργασίας ε, για την καταπολέμηση της φτώχειας και του κοινωνικού αποκλεισμού γιατί μιλήσαμε για την ανάγκη εδαφικής και κοινωνικής συνοχής. Στη διάρκεια της Προεδρίας θα οργανώσουμε και την ετήσια διάσκεψη της Ευρωπαϊκής ε, Πλατφόρμας Συνεργασίας κατά της Φτώχειας, όπως σας είπα, και του κοινωνικού αποκλεισμού. Στόχος ε, της διάσκεψης αυτής, ε, του συνεδρίου αυτού, είναι μια επισκόπηση των πρόοδων σε ό,τι αφορά την υλοποίηση των κοινωνικών στόχων της στρατηγικής του 2020 και σίγουρα η καταπολέμηση της φτώχειας είναι πολύ σημαντικό θέμα και μια παρακολούθηση, η επισκόπηση μάλλον των εθνικών στρατηγικών καταπολέμησης της φτώχειας. Θα προσπαθήσουμε να υποβάλουμε και συγκεκριμένες προτάσεις για το θέμα αυτό. Πολλές από εσά μιλήσατε για την αναπαραγωγική υγεία, για τη διάκριση λόγω Όλα αυτά τα θέματα φυσικά αντιμετωπίζονται στην εθνική νομοθεσία. Έχουμε σχετικές νομοθετικές διατάξεις. Δεν είναι όλα αυτά τα θέματα λιμένα σε ευρωπαϊκό επίπεδο. Γι' αυτό θα ήθελα να σας προσκαλέσω θερμά στη διάσκεψη, γιατί εκεί θα γίνουν εκτενείς συζητήσει και θα σας παρουσιάσουμε τις εθνικές μας διατάξεις για τα θέματα αυτά. Δεν ξέρω, κύριε Πρόεδρε, μακρηγόρησα. Ευχαριστώ. Και τώρα η κυρία Ρατισεύσκα έχει το λόγο. Ευχαριστώ. Εγώ πόσα λεπτά έχω. Six. Ah. <laughs> Έξι. Καλώς. Θα προσπαθήσω να ομαδοποιήσω τις ε, ερωτήσεις. Δεν θα απαντήσω μεμονωμένα στην κάθε ευρωβουλευτή, γιατί πραγματικά έχω ελάχιστο χρόνο στη διάθεσή μου. Αναφέρθηκαν τα αναπαραγωγικά δικαιώματα και το θέμα των αμβλώσεων. Πολλές παρατηρήσεις έγινε αυτό. Το θέμα των αμβλώσεων και των αναπαραγωγικών δικαιωμάτων είναι εθνική αρμοδιότητα και εμείς έχουμε αρκετά αυστηρό δίκαιο όντως στην Πολωνία και έγιναν συζητήσεις γιατί ζητήθηκε να γίνουν ακόμη πιο αυστηρέ αυτές οι νομοθετικέ διατάξεις. Έγινε σφοδρή συζήτηση γι' αυτό. Το σχέδιο αυτό είναι σχέδιο για τους πολίτες και σε ευρωπαϊκό επίπεδο. Ε, οι πολίτες έχουν δικαίωμα να υποβάλουν τις προτάσεις τους στη, η πολωνική νομοθεσία προβλέπει ότι 100.000 πολίτε ε, με υπογραφές μπορούν να υποβάλουν νομοθετική πρόταση. Στην Πολωνία είχαμε 500.000 υπογραφές και έγινε σχετική συζήτηση στην Πολωνική Βουλή. Επειδή ε, ε, είναι πολύ συγκινησιακά φορτισμένο αυτό το θέμα γιατί έχει και διοντολογικό και ηθικό αντίκτυπο και πτυχές Και μάλιστα τον Οκτώβριο, στις 9 Οκτωβρίου θα γίνουν οι βολευτικέ εκλογέ. Οπότε κατά πάσα πιθανότητα το θέμα αυτό δεν ε, θα ολοκληρωθεί, δεν θα δοθεί μια νομική λύση. Σίγουρα θα συνεχιστούν οι συζητήσει ε, και στην επόμενη κοινοβουλευτική θητεία. Γιατί θα δείτε ότι έγιναν προτάσεις ε, και για την ε, προαιρετική άμβλωση. Ήταν ευρύ το φάσμα της συζήτησης. Πάντως ε, δεν είναι και πολύ κακή κατάσταση για τα αναπαραγωγικά δικαιώματα στην Πολωνία, γιατί κάθε γυναίκα έχει δικαίωμα για κοινωνική ασφάλιση και μάλιστα κοινωνική ασφάλιση που τη χρηματοδοτεί το κράτος. Κάθε, ακόμη και δεν εργάζεται, κάθε γυναίκα έγκυος έχει δικαίωμα στην στην ε, υγειονομική περίθαλψη. Και μάλιστα θέλουμε μερικές φορές ε, ατομικέ προσκλήσεις στις γυναίκες για να κάνουν τις εξετάσεις που χρειάζονται και μερικές φορές οι ίδιες δεν θέλουν, ενώ δεν υπάρχει πρόβλημα οικονομικό. Και τους δίνουμε συγκεκριμένα ραντεβού. εμείς ε, κυνηγάμε κατά κάποιο τρόπο τις γυναίκες για να κάνουν τις εξετάσεις και δυστυχώ οι γυναίκε αμελούν την ε, πραγματοποίηση των εξετάσεων και πραγματικά έχουμε αρκετούς θανάτους από καρκίνο του μαστού και καρκίνο τραχύλου της Μήτρα, ιδιαίτερα σε μικρούς δήμου και κοινότητε, Γι' αυτό και προσπαθούμε να ευαισθητοποιήσουμε τις γυναίκες για να κάνουν πιο τακτικά τις ιατρικές εξετάσεις. Θα ήθελα επίσης να σας διαβεβαιώσω ότι όλες ε, οι νομικές διατάξεις ε, της Πολωνίας εξασφαλίζουν πλήρη δικαιώματα για, τις, ε, για την ομάδα GLBT, δηλαδή ομοφιλοφίλους άνδρες και γυναίκες ε, ε, και φιλομεταβατικούς. Δεν έχουμε διακριτικές μεταχειρήσεις για τέτοιους λόγους, για να ο Και μάλιστα κάποιος που θεωρεί ότι είναι θύμα διακριτικής μεταχείρισης μπορεί να διεκδικήσει αποζημίωση. Και μάλιστα εδώ έχουμε αντιστροφή του βάρου απόδειξη. Δηλαδή σε περίπτωση που κάποιο ε, θεωρεί ότι είναι θύμα, δεν πρέπει να αποδείξει ότι είναι θύμα, αλλά ο αυτούργό τη διάκριση θα πρέπει να αποδείξει ότι δεν ε, ε, διέπραξε διακριτική μεταχείριση. Οπότε οι ομοφυλόφιλοι άνδρε και γυναίκε και φιλομεταβατικοί και αμφωτεροφιλόφιλοι δεν υφίσταται διακριτική μεταχείριση και ούτε έχουμε προβλήματα με τις gay pride που οργανώνονται και με την υποστήριξη μη κυβερνητικών οργανώσεων. Τώρα, σε ό,τι αφορά την ύπαρξη όχι πολωνικού προγράμματος για τα θέματα ισότητας και ιδιαίτερα ισότητας των φύλων. Μέχρι στιγμής δεν είχαμε ένα ευρύ πρόγραμμα, αλλά νομικά προβλέπεται, νομοθετικά προβλέπεται και θα υλοποιηθεί. Έχουμε ήδη ξεκινήσει εργασίες και μάλιστα στα πλαίσια του κυβερνητικού προγράμματος και στα πλαίσια της χρηστής διακυβέρνησης ε, έχουμε 400 ε, ε, υπαλλήλου από πολλούς δήμους και κοινότητες και στα πλαίσια αυτού του σχεδίου θα εκπονήσουμε μια στρατηγική με βάση ευρύτατες μελέτες και έρευνες που έχουν γίνει και τώρα και προηγουμένως και θα ήθελα να σας πω ότι στα πλαίσια του σχεδίου αυτού, για πρώτη φορά στην ιστορία της Πολωνίας, η κυβέρνηση έκανε έρευνες και μελέτες για τη διακριτική μεταχείριση της ομάδας των ομοφιλοφίλων, φιλομεταβατικών και φωτεροφιλόφίλων με κρατικά κονδύλια. Για πρώτη φορά έγιναν μελέτες και έρευνες για το θέμα αυτό με συμμετοχή ακαδημαϊκών κύκλων και καθηγητών πανεπιστημίων, άρα εξασφαλίζεται η αμεροληψία και με βάση τα απορίσματα αυτών των μελετών θα καταρτιστεί κυβερνητικό σχέδιο για την ίση μεταχείριση και πάταξη των διακρίσεων για λόγους φύλου αλλά και για λόγους γενετήσιου προστρατορισμού. Και έτσι θα υπάρξει οριζόντια λήψη υπόψη το θέματος αυτού στα 17 Υπουργεία. Το θέμα της ισότητας των φύλων είναι πολύ σημαντικό και θα γίνουν μελέτες για το τι ρυθμίσει χρειάζονται για να βελτιωθεί η κατάσταση, αλλά και για το θέμα των ε, δικαιωμάτων των ε, ομοφιλοφίλων και φιλομεταβατικών γίνονται πλήρω σεβαστά τα δικαιώματά τους. Τώρα, καλύτερη αμοιβή των γυναικών ή εξίσωση των μισθών, εξίσωση των συντάξεων, γιατί αυτή τη στιγμή υπάρχουν συντάξει πείνα, ειδικά για τι γυναίκε. Και οι γυναίκε μερικέ φορέ ε, οι συνταξιούχε, Έχουμε για πρώτη φορά ένα πορτάλ στο διαδίκτυο, μια διαδικτυακή πύλη, στην οποία συμμετέχουν οι μεγαλύτερες επιχειρήσεις, ε, ενώσεις δικαιωμάτων ε, ε, των οικογενειών και το οικονομικό επιμελητήριο και γίνονται καταγγελίες γιατί Χάρη στα προγράμματα αυτά θα, γίνουν, θα γίνει καλύτερη ενημέρωση, θα γίνει καλύτερη ενημέρωση, ανταλλαγή πρακτικών για να γνωρίζουν όλοι τα δικαιώματά τους και να μπορούν να τα διεκδικούν. Και το θέμα της καταπολέμησης της βίας ε, κατά των γυναικών είναι πραγματικά μία μάστιγα. Θα συνεχίσουμε λοιπόν την προσπάθεια ε, θα έχουμε την 6η Δεκεμβρίου την ε, μάχη των ανδρών κατά της βίας κατά των γυναικών. Δηλαδή θα πρέπει να αναμίξουμε και τους άνδρες, ε, να εκφράσουν τη γνώμη τους και να πούν ότι δεν επιτρέπεται βία κατά των γυναικών. Η βία δεν είναι τρόπος ε, συζήτησης, ούτε τρόπος διαλόγου, ούτε στην οικογένεια, ούτε στην, στον εργασιακό χώρο, ούτε πουθενά. Και θέλουμε συμμάχους στη διοργάνωση αυτή, στη 6 Δεκεμβρίου, αυτή την πανευρωπαϊκή εκστρατεία κατά της βίας. Και κάτι ακόμη. Στην Πολωνία έχουμε πολλές εκκλησίες και η εκκλησία είναι στοιχείο της καθημερινότητας πολλών Πολωνών. Γιατί πολλές φορές μιλούμε για την βία κατά των γυναικών, για την κακή μεταχείριση επιχειρήσεις, για, την απο... τον αποκλεισμό των αναπήρων, την περιθωριοποίηση των ηλικιωμένων. Έχω μία ομάδα διαθρησκευτική με συμμετοχή πολλών εκκλησιών και καταλήξαμε σε μια συμφωνία και στις 25 Νοεμβρίου θα έχουμε την Παγκόσμια ημέρα πολέμηση της βίας ε, εις βάρος των γυναικών και όλες οι εκκλησίες θα συμμετέχουν σε αυτήν την ε, εκστρατεία και οι τρεις εκκλησίες, και η Καθολική και η Ορθόδοξη και η Λουθυρανική, αλλά ακόμη και η Μουσουλμανική κοινότητα και η Εβραϊκή κοινότητα θα συμμετέχει. Και ελπίζω κάθε χρονιά να βελτιώνεται η συμμετοχή, ώστε να αυξηθεί η συνειδητοποίηση και να περιοριστεί η ενδοοικογενειακή βία. Επίσης, ε, θέλουμε έκκληση, να απευθύνουμε έκκληση προς τους εργοδότες να προσλαμβάνουν γυναίκες, γιατί οι γυναίκες είναι μορφωμένες, καταρτισμένες και έχει συμφέρον ο εργοδότης να προσλαμβάνει γυναίκες. Είναι προς το συμφέρον του, είναι καλές ε, εργαζόμενες και η απόδοση θα είναι πολύ μεγαλύτερη. Και Έχουμε τις νομοθετικές διατάξεις, αλλά μερικές φορές άλλο η νομοθετική διάταξη και άλλο η πρακτική εφαρμογή. Εμείς θέλουμε να κινητοποιήσουμε κάθε μηχανισμό ώστε να εφαρμόσουμε και στην πράξη τις νομοθετικές διατάξεις που ήδη υπάρχουν και κατοχυρώνουν αυτά τα δικαιώματα. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ. Λυπούμε που δεν έχουμε επαρκή χρόνο αλλά υπήρχε πολύ ενδιαφέρον, σας απευθύνθηκαν πολλές ερωτήσεις, προσβλέπουμε στην συνεργασία με την Προεδρία και σας εύχομαι καλή επιτυχία ευχαριστώντας σας πάρα πολύ. Παρακαλώ, θα συνεχίσουμε τώρα. Ας περάσουμε τώρα στο στοιχείο 5 της ημερήσιας διάταξης. Ανακοινώσει σχετικά με ε, τη συνάντηση των συντονιστών, τα αποτελέσματα ε, των αποφάσεων των συντονιστών στις 27 Ιουνίου. Θα βρείτε στα αρχεία σας ε, τα πρακτικά αυτά. Σας ε, έχουν διανεμηθεί και έχουν διανεμηθεί και στα μέλη του Κοινοβουλίου. Εάν δεν έχετε αντιρρήσεις θα τις εγκρίνουμε. Η κυρία Μπάουερ ζήτησε το λόγο. Ευχαριστώ πολύ. Ήθελα να κάνω έκκληση προς τους συναδέλφους μου να επαναφέρουν το ζήτημα του συνόλου κανόνων για τα θύματα στην ε, συνεδρίαση συντονιστών επειδή του ζήτησαν να συσχετίσουν τις ε, διαπραγματεύσεις με μια πρόταση κανονισμού που θα αποσκοπεί στην ολοκλήρηση του αμοιβαίου εργαλείου για τα προστατευτικά μέτρα, για ποινικά θέματα και για την διασφάλιση του ότι όλα τα μέτρα προστασίας θα υποφελούνται από ένα μηχανισμό στήριξης. Δεν έγινε κατανοητό και συσχετίστηκε με τα δικαιώματα των θυμάτων απευθείας. Πιστεύω ότι δεν ήταν αρμόζουσα μια τέτοια απόφαση. Η πρότασή μου για το συσχετισμό με τα νομοθετικά μέσα, νομοθετικών μέσων που είναι αλληλοσυμπληρωματικά. Έγινε απόφαση για συσχετισμό δύο άλλων νομοθετικών μέσων. Θα ήθελα λοιπόν να σας ζητήσω να το ξαναδώσουμε στη συνάντηση των συντονιστών και να επανεξεταστεί η απόφαση αυτή. Ευχαριστώ κυρία Πάουερ. Υπάρχει λοιπόν μια αντίρρηση. Αντίρρηση όσον αφορά τα αποτελέσματα της συνάντησης των συντονιστών στις 27 ε, Ιουνίου. Θα ήθελα να κάνω την ακόλουθη παρατήρηση. Δεν νομίζω ότι υπήρχε παρανόηση. Ήταν μια σαφής απόφαση που ελήφθη από τους συντονιστές. Ε, δεν πρόκειται για παρανόηση καθόλου. Αν έχετε αντίρρηση για αυτή την απόφαση, τότε η ρόλη είναι πολύ σαφής. Σε αυτή την περίπτωση η Επιτροπή θα πρέπει να ψηφίσει για αυτήν τη συγκεκριμένη απόφαση, την αμφισβητούμενη απόφαση και αν η πλειοψηφία αντιτίθεται στην απόφαση, τότε το ζήτημα θα παραπεμφθεί σε μια άλλη συνεδρίαση των συντονιστών κάποια στιγμή στο μέλλον. Αυτό είναι ο κανόνα. Συνεπώ, θέτω αυτό το ζήτημα σε ψηφοφορία Αναφέρομαι στα πρακτικά της συνάντησης των συντονιστών της 22ης Ιουνίου. Ήταν το ε, σημείο που αφορά το πακέτο για τα θύματα, το σύνολο μέτρων για τα θύματα. Όσοι από εσάς πιστεύετε ότι η απόφαση που ελήφθη στη συνεδρίαση των συντονιστών θα πρέπει να είναι έγκυρη, να ισχύει, σηκώστε τα χέρια σας τώρα. ευχαριστώ όσοι υποστηρίζετε την πρόταση της κυρίας Μπάουερ, έχετε αντίρρηση προς αυτή την απόφαση, σηκώστε τα χέρια σας. Ευχαριστώ πολύ ψηφίστηκε λιπτό το ζήτημα. Το αποτέλεσμα είναι ότι οι 13 ε, βουλευτές ψήφισαν υπέρ της διατήρησης της απόφασης που έλαβαν οι συντονιστές στις 22 Ιουνίου 10 ψήφισαν κατά συνεπώς η Επιτροπή έχει αποφασίσει ότι η απόφαση των συντονιστών της 22 Ιουνίου θα ισχύσει. Ας προχωρήσουμε τώρα με την ημερήσια διάταξη. Ας ξεκινήσουμε με τις ψηφοφορίες. Θα ξεκινήσουμε με το στοιχείο της κυρίας Σιγκλιεύσκα. ημερήσια διαταξή για τις νέες δεξιότητες και θέσεις εργασίας. Έχετε το λόγο. Ευχαριστώ ξέρω ότι έχουμε μείνει πίσω στο χρόνο. Θα ήθελα εν συντομία να ευχαριστήσω θερμά όλους τους και οδησηγητές για τις τροπολογίες τους. Να ευχαριστήσω τους βουλευτές και τις πολιτικές ομάδες ε, και να εκφράσω την ικανοποίησή μου για τις συμβαστικές λύσεις που βρήκαμε. Ελπίζω να εγκριθεί η έκθεση όπως ε, διαμορφώθηκε στην Επιτροπή Κοινωνικών Υποθέσεων. Ευχαριστώ πολύ. Έτσι, περνάμε στην ψηφοφορία. Ξεκινάμε με το συμβιβασμό 2, υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται συμβιβασμό 3, κατά, αποχή, συμβιβαστική 4, υπέρ, κατά, αποχές εγκρίθηκε. Περνάμε στη συμβιβαστική 5 υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίθηκε στην 6 υπέρ. Κατά. Αποχή εγκρίθηκε 7 υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίθηκε 8 υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίθηκε. Και τώρα έχουμε τη συμβιβαστική 9 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται τροπολογία 11 υπέρ κατά αποχές εγκρίθηκε έχουμε ξεκινήσει την ψηφοφορία κλείνει η ψηφοφορία απορρίπτεται Έχετε κάρτα και μάλιστα και ψηφίζετε. Συνεπώς απορρίπτεται. Ψηφίζετε υπέρ, αλλά παρόλα αυτά απορρίπτεται. Μάλιστα. Περνάμε στην τροπολογία 12 υπέρ, κατά, αποχές, απορρίπτεται, 13 υπέρ, κατά, αποχές ε, απορρίπτεται 14 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται 15 ανοίγει ψηφοφορία λίγη ψηφοφορία Έχει κλείσει η ψηφοφορία, είναι υπέρ 16, υπέρ 14 κατά. Τώρα έχουμε... Την υπολογίσαμε. Την υπολογίσαμε την κυρία Κώστα, έχει ψηφίσει. τροπολογία 14 έχει εγκριθεί. Περνάμε στην τροπολογία 18. Υπέρ για την 18. Κατά. Αποχές απορρίπτεται. 19. Υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. 27. Υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. ψηφίσουμε για την 27. Ξεκινάει η ψηφοφορία. Περισσεύει ένας από τους σοσιαλιστές. Τώρα είμαστε εντάξει. Κλείνει η ψηφοφορία, εγκρίνεται. 29 υπέρ για το δεύτερο μέρος μόνο 29 το δεύτερο μέρος υπέρ για το τροπολογία 29 το δεύτερο μέρος υπέρ το ΕΛΚ ζήτησε να ψηφιστεί το δεύτερο μέρος, παρακαλώ το 29, το δεύτερο μέρος υπέρ, κατά, αποχές, νομίζω εγκρίθηκε. Ε, ανοίγουμε την ψηφοφορία για το δεύτερο μέρος του 29. Λίγη ψηφοφορία. Εγκρίνεται. 32. Υπέρ κατά καταπίπτει οπότε περνάμε στην 36 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται 35 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται 37 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται 38 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 40 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 41 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 40 ας ελέγξουμε το 41 ξεκινάει η ψηφοφορία λίγη ψηφοφορία εγκρίνεται 42 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται 43 να ελέγξουμε την 42 ψηφίζουμε αρχίζει ψηφοφορία για την 42 λίγη ψηφοφορία απορρίπτεται 43 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Να ελέγξουμε και για την τροπολογία 43 ανοίγει η ψηφοφορία. Λίγη η ψηφοφορία. Εγκρίνεται. 52 υπέρ. Κατά. Αποχή. Εγκρίνεται. 53 υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. Και τώρα περνάμε στις τροπολογίες ε, στη συμβιβαστική 1 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Ε, τροπολογία 1 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. 2 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Τροπολογία 4 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται. Τροπολογία 7 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται. Τροπολογία 8 να ελέγξουμε την 7 ξεκινάει η ψηφοφορία. Λίγη ψηφοφορία. Εγκρίνεται. 16 ε, υπέρ και 14 κατά ψήφισαν. 8 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Να ελέγξουμε την 8, ξεκινάμε την ψηφοφορία. Λίγη ψηφοφορία. Ε, απορρίπτεται τελικά 15 προς 15. και εσείς ψηφίσατε όχι, απορρίπτεται. Ε, αριθμός 9 υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. 10 υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. Και τώρα έχουμε την τελική ψηφοφορία, ξεκινάει η ψηφοφορία. Λίγη ψηφοφορία. Εγκρίνεται. Συγχαρητήρια. Can you take off the because it makes noise for Yeah, yeah. Ας προχωρήσουμε με το επόμενη ψηφοφορία αφορά την έκθεση για την κατάσταση των γυναικών που πλησιάζουν την ηλικία συνταξιοδότηση. Θα δώσω το λόγο στην κυρία Μπάουερ ώστε να κάνει μερικά σχόλια πριν ξεκινήσουμε την ψηφοφορία. Κυρία Μπάουερ, παρακαλώ. Κυρία Μπάουερ, αν θέλετε να πείτε κάτι πριν ξεκινήσουμε την ψηφοφορία σχετικά με την ε, έκθεσή σας. Κυρία Μπάουερ, έχετε το λόγο. Ευχαριστώ. Θέλω να ευχαριστήσω όλους τους σκιώδεις εισηγητές και όλους αυτούς οι οποίοι ε, βελτίωσαν το σχέδιο της εκθέσεως μέσω των τροπολογιών. Μπορέσαμε να επιτύχουμε επιτυχείς ε, συμβιβαστικές λύσεις. Ευχαριστώ κυρία Μπάουερ. Ε, ξεκινάμε καταρχήν με την τροπολογία 21. Υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. 23. Υπέρ, κατά, αποχές, απορρίπτεται. 24. Υπέρ. Να ελέγξουμε την 23 με ηλεκτρονική ψηφοφορία. έληξε. Και απερίφθη παρόλα αυτά. Τώρα όσον αφορά την 24 υπέρ, κατά, αποχές εγκρίνεται 25 υπέρ, κατά, αποχές εγκρίνεται 26 υπέρ, κατά, αποχές εγκρίνεται. Τώρα έχουμε τη συμβιβαστική 4 και υπάρχει μία προφορική τροπολογία σχετικά με την τέταρτη συμβιβαστική. για να αλλάξουμε τους όρους financial liability του healthcare και να αλλάξει να είναι affordability of healthcare. Έχει κάποιος αντίρρηση? Όχι τότε μπορούμε να ψηφίσουμε τη συμβιβαστική τροπολογία 4 με αυτή την προφορική τροπολογία. Υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. 31 ε, υπέρ, κατά, αποχές, απορρίπτεται. 33 ε, υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. Συμβιβαστική 5 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. 35 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. 36 υπέρ κατά αποχές Συμβιβαστική 6 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Ε, η συμβιβαστική 7 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται.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 65 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται συμβιβαστική 11 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 66 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 68 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 69 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 70 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 71 σε δύο τμήματα το πρώτο τμήμα ποιος είναι υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται δεύτερο τμήμα του, της 71 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 72 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 73 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται και τώρα ερχόμαστε στην 74 υπέρ έχουμε όμως και μία την ε, προφορική τροπολογία η ίδια με την συμβιβαστική 4 ε, να αλλάξουμε το financial το affordability of Health healthcare, σκέτο affordability, υπέρ κατά αποχές ε, εγκρίνεται, 75 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται, 76 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται, 77 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται, 78 υπέρ κατά αποχές ε, απορρίπτεται 79 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 80 ε, ε, υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 81 ε, υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 72 καταπίπτει 83 υπέρ κατά Νομίζω ότι πρέπει να κάνουμε ηλεκτρονικό έλεγχο. Νομίζω ότι απερίφθη, αλλά ας ελέγξουμε. Λίγη ψηφοφορία και όντως ε, απερίφθη. 84, τέσσερα υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 85 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 86 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 87 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται συμβιβαστική 12 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται και τώρα ερχόμαστε στην 90 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται 91 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 92 σε δύο τμήματα πάλι το πρώτο μέρος υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται δεύτερο τμήμα της 92 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 93 Ας ελέγξουμε για το δεύτερο τμήμα της τροπολογίας 92. Λίγη ψηφοφορία και απερίφθη. Το 93 υπέρ κατά αποχές ε, εγκρίνεται και 94 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Τροπολογία 2 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. 3 υπέρ κατά αποχές ε, απορρίπτεται. 4 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. 5 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 6 σε 2 τμήματα το πρώτο τμήμα ποιος είναι υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται δεύτερο τμήμα υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται συμβιβαστική 1 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 9 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται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 19 υπέρ κατά απορρίπτεται και τέλος συμβιβαστική 3 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται και τελική ψηφοφορία ξεκινά λίγη εγκρίθηκε και συγχαίρουμε την κυρία Μπάουερ. Τώρα... Τώρα θα... Τώρα θα περάσουμε στο επόμενο στοιχείο το οποίο, για το οποίο επίσης θα ψηφίσουμε. Πρόκειται για μια γνωμοδότηση προς την Επιτροπή ΙΤΡΕ σχετικά με την πράσινο βιβλό με τίτλο «Από τις προκλήσεις της ευκαιρίες προς ένα κοινό πλαίσιο στρατηγικής για τη χρηματοδότηση της έρευνας και της καινοτομίας στην Ευρωπαϊκή Ένωση». Η συντακτρία για τις νομοδότησης ήταν η Κύπρια Μπρίτα Τόμσεν για την Επιτροπή μας. Δεν ξέρω αν θα ήθελα να κάνει κάποια σχόλια πριν ξεκινήσουμε. Έχετε το λόγο, όχι. Μπορούμε λοιπόν να ξεκινήσουμε την ψηφοφορία. Η κυρία Μπάουερ θέλει να πει κάτι. Μπορούμε να ψηφίσουμε ε, μαζικά για όλα, όλες τις τροπολογίες. Υπάρχει αντίρρηση γι' αυτό σχετικά με την μαζική, πρόταση μαζικής ψηφοφορίας. Ναι, υπάρχει αντίρρηση. Θα χρειαστεί λοιπόν να ψηφίσουμε κανονικά.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 Παίρναμε στην τροπολογία 6 υπέρ, κατά, αποχές εγκρίνεται, 7 υπέρ, κατά, αποχές εγκρίνεται, η 11 ε, υπέρ, κατά, αποχές εγκρίνεται, 12 υπέρ, κατά, αποχές εγκρίνεται, 13 υπέρ, κατά, αποχές εγκρίνεται, 14 υπέρ, κατά, αποχές εγκρίνεται 19 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 20 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 23 υπέρ και 24 ψηφίζουμε για την 23 και την 24 υπέρ κατά απορρίπτεται. Η επόμενη είναι η τροπολογία 30. Υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. 32 υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. Η 1 υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. 2 υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. 3 υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. Και τελική ψηφοφορία ξεκινάει. Λίγη η ψηφοφορία. Εγκρίνεται. Λοιπόν, συγχαρητήρια κυρία Τόμσεν. And the next one. Nästa ärende vi ska rösta om, det är ett... Το επόμενο στοιχείο για ψηφοφορία είναι μια γνωμοδότηση που υποβάλλουμε στην Επιτροπή Ανάπτυξη. Έχει πολύ μεγάλο τίτλο. Σχέδιο γνωμοδότηση σχετικά με το ρόλο τη ιδιοκτησία, των δικαιωμάτων ιδιοκτησία και την παραγωγή πλούτου για την εξάλληψη τη φτώχεια και την πρόθεση της βιώσιμης ανάπτυξης στις αναπτυσσόμενες χώρε. Συντάκτρια είναι η κυρία Κώστα και θα ήθελα να της δώσω το λόγο. Θέλω να ευχαριστήσω τους συναδέλφους όλων των ομάδων που συνέβαλαν στη σύνταξη. Σήμερα έλαβε χώρα ένα καταπληκτικό σεμινάριο με ορισμένους συναδέλφους της Επιτροπής Γεωργίας και Ανάπτυξης και εκεί προέκυψε ότι η προοπτική πρόσβαση σε πορούς όπως το νερό θα είναι ένα μεγάλο θέμα για το οποίο θα πρέπει να αποφασίσει το Κοινοβούλιο. Είναι ενδιαφέρον λοιπόν να συνεχίσουμε σε αυτή την Επιτροπή για τις Γυναίκες για τα... να συζητάμε για τα ζητήματα ανάπτυξης, ε, γεωργίας και ε, πόρων. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ κυρία Κώστα. Ας ξεκινήσουμε με την ψηφοφορία. Συμβιβαστική ένα υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. 11, καταπίπτει. Έτσι περνάμε στην τροπολογία 15 υπέρ κατά αποχές εγκρινέται 16 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται. Συμβαστική 2 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται και τώρα 23 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Συμβαστική 3 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Συμβιβαστική 4 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 28 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 29 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 30 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 34 ε, συμβαστική 5 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται και περνάμε στην πισωσελίδα, στην τροπολογία 1 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. 6 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Τροπολογία 5 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. 6 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. 7 συμβιβαστική υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. 10 υπέρ κατά απορρίπτεται. Ας το ελέγξουμε την τροπολογία 10. Ανοίγει ψηφοφορία. Κλείνει ψηφοφορία. Απορρίπτεται. Τελική ψηφοφορία. Κλείνει η ψηφοφορία. Εγκρίνεται. Συγχαρητήρια στην κυρία Κώστα. Och ναι. det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 wanted to say, and it's a little bit going to a different direction, so I don't think it's appropriate in this case. Tack Mrs Pavanova. Då röstar vi om ändringsförslag nummer 11 utan något muntligt ändringsförslag. Nummer 11, vote in favor. Against, abstention, adopted. Number 12 in favor. Against, abstention rejected. Let's check. We check. The vote is opened. Ηλεκτρονικός έλεγχος ξεκινάει, λίγη και απερίφθη. Συμβιβαστική 4 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Πάμε τώρα στην 14 υπέρ κατά αποχές ε, απορρίπτεται. Ας ελέγξουμε τη 14. Λίγη η ψηφοφορία. Απερίψη. 17 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. 18 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. 20 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. 19 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. 21 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. 22 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται. 23 σε τρία τμήματα, πρώτο τμήμα 25 μάλλον σε τρία τμήματα. Πρώτο τμήμα υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. Δεύτερο τμήμα υπέρ, κατά, αποχές. Ας ελέγξουμε το δεύτερο τμήμα της 25 ξεκινάει. Λίγη. Απερίφθη. 25. Τρίτο τμήμα. Προφορική τροπολογία από την κυρία Τζαμπόσκα. Έχει κάποιο αντίρρηση σχετικά με την, το τρίτο μέρος της τροπολογίας 25 με προφορική τροπολογία έχουμε όμως α, α, α, ε, αντίρρηση άρα ψηφίζουμε την αρχική τροπολογία υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 26 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 27 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 28 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 29 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 1 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Θα ελέγξουμε την 1 ε, ηλεκτρονικά. Ξεκινάει η ψηφοφορία, λίγη ψηφοφορία και ενεκρίθη. Συμβιβαστική 1 ε, υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. 4 ε, υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. 5 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται και τώρα υπάρχει η τελική ψηφοφορία ηλεκτρονικά, ξεκινά, λίγη και ενεκρίθη. Θέλω να συγχαρώ την κυρία Κορνέλισεν. Λοιπόν, ευχαριστώ. Ευχαριστώ όλους τους συναδέλφους γιατί πήγαν πολύ καλά οι ψηφοφορίες σήμερα και μπορούμε να προχωρήσουμε στο επόμενο θέμα της ημερησίας διατάξεως. Ας περιμένουμε ένα-δυο λεπτά ώστε να μπορούν να μπουν όσοι θέλουν πριν φτάσουμε στο επόμενο θέμα. now Nu börjar vi igen. και προχωράμε στο επόμενο θέμα. Εάν έχετε κάτι να συζητήσετε, παρακαλώ εκτός εθούσης, γιατί ξαναξεκίνησαν οι εργασίες μας. Το επόμενο θέμα είναι η Ευρωπαϊκή ε, πολιτική, η συμβολή των πολιτικών οι οποίες προωθούν την ισότητα ανδρών και γυναικών στην καταπολέμηση της εγκληματικότητας των νέων και η συγγήτρια είναι η κυρία Ζαμπόρσκα. Την παρακαλώ λοιπόν να παρουσιάσει το θέμα αυτό για να μπορέσουμε να συζητήσουμε και την έκθεση. Ευχαριστώ, κυρία Πρόεδρε. Θα ήθελα να σας ευχαριστήσω διότι μπορέσατε κάπως να προσαρμόσετε την ημερήσια διάταξη καθότι υπάρχουν σοβαροί λόγοι για τους οποίους αύριο δεν θα μπορέσω να συμμετάσχω ή στην συνεδρίαση της Επιτροπής και ερχόμαστε τώρα στην επεξεργασμένη έκθεση σχετικά με τη συμβολή ορισμένων ευρωπαϊκών πολιτικών στην ισότητα ανδρών γυναικών και στην καταπολέμηση της εγκληματικότητας των νέων. Θα ήθελα λοιπόν να μην αναφερθώ εδώ σε συγκεκριμένα θέματα τα οποία έχουμε θίξει στο παρελθόν και γι' αυτό στο κείμενο αυτό πρέπει να τονίσουμε ότι υπάρχουν πολλές πολιτικές οι οποίες ε, επικεντρώνονται στην ισότητα των φύλων και που μπορούν να συμβάλλουν στην καταπολέμηση της εγκληματικότητας των νέων όχι μόνο σχετικά με την ισότητα των ευκαιριών, αλλά με συντονισμό της ε, οικογενειακής ε, ε, ζωής με την επαγγελματική και των επιπτώσεων στον κοινωνικό και οικονομικό τομέα. Στην έκθεσή μου προσπάθησα να αναφέρω αυτά τα θέματα και ενδεχομένως θα μπορούσε κανείς να έχει επεκταθεί και περαιτέρω αλλά ε, επειδή υπάρχουν ορισμένοι κανονισμοί στο ε, καταστατικό δεν έχουμε μεγάλη ευελιξία είναι όμως δυνατόν στα πλαίσια της ε, εργασίες μας να περιοριστούμε στα ουσιαστικά. Όπως και στην πρώτη έκθεση ε, υπήρχαν ε, σαν σημείο εκκινήσεως ορισμένα ε, σημαντικά έγγραφα της Ευρωπαϊκής Ενώσεως. Συνεργάστηκα και με ορισμένες διεθνείς οργανώσεις οι οποίες έχουν παρέμβει. Πρόκειται για τον ΟΗΕ, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, την Κοινωνική και Οικονομική Επιτροπή για το Συμβούλιο της Ευρώπης ή για την Παγκόσμια Τράπεζα. Και προσπάθησα να διατυπώσω κατά αυτόν τον τρόπο την έκθεση ώστε να μην επηρεαστώ από τις μελέτες που έχουν κατακτηστεί από μη κυβερνητικέ οργανώσεις ή άλλους εξωτερικούς παράγοντες. Ήθελα όμως ε, να αποκλείσω τις πολύ αμφιλεγόμενες απόψεις ε, και όσον αφορά την πολιτική γραμμή η οποία είναι σημαντική για το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο πρέπει να πω ότι όταν πρώτο συζητήσαμε το θέμα αυτό υπήρξαν παρατηρήσεις από πολλούς συναδέλφους και αυτό που μας απασχόλησε τότε ήταν ότι στην έκθεση αυτή δεν είχε οριστεί επαρκώς η εγκληματικότητα. Προσπάθησα λοιπόν στα επίσημα έγγραφα να αναφερθώ ως έναν ορισμό και ο μόνο ε, αποκλεισμός ε, ορισμένων εγγράφων όπως ελάχιστες προδιαγραφές είχε περιληφθεί σε ένα έγγραφο του ΟΗΕ και γι' αυτό προχώρησα βάσει αυτών των κριτηρίων. Δηλαδή και εγώ εργάστηκα σύμφωνα με τους ορισμούς του ΟΗΕ με ε, τον ορισμό για τον ε, νέο, για τον ε, ενήλικα, για τον ορισμό μίας αξιόπινης ή εγκληματικής πράξης ε, και θεωρώ ότι ένας ε, νέος ε, εγκληματίας είναι κάποιος ο οποίος έχει διαπράξει μία αξιόπινη πράξη. Βεβαίως δεν είναι μόνο το θέμα των ανηλίκων και των νέων που διαπράττουν αξιόπινες πράξεις. Ε, ε, υπάρχουν αξιόπινες ε, πράξεις και βία που εξασκείται όχι μόνο προς τους ενήλικες αλλά και προς αγόρια και κορίτσια. Υπάρχουν ποινικά δικήματα, υπάρχουν παραβιάσεις και πολλές φορές οι πράξεις αυτές υποκινούνται από τον αλκοολισμό, την ε, αναζήτηση ναρκωτικών ή τη χρήση ναρκωτικών. Γι' αυτό και στην περίπλοκη παρακολούθηση και αξιολόγηση του θέματος θα πρέπει όλα αυτά τα θέματα να ληφθούν υπόψη εφόσον μπορούν να οδηγήσουν τους νέους προς, μια, ε, προς τη διάπραξη αξιόπινης πράξης η Οικονομική και Κοινωνική Επιτροπή έχει την, ε, πιο τον πιο πλήρη ορισμό συμπεριλαμβάνοντας κοινωνικούς παράγοντες και για τους ανήλικες και για τους παράγοντες που μπορεί να επηρεάσουν την δραστηριότητά τους. Εγώ προσπάθησα απλώς να απαριθμίσω αυτή την ε, ε, δύσκολη κατάσταση η οποία μπορεί να οδηγήσει σε εγκληματικές πράξεις. Επιπλέον, προσπάθησα να τονίσω την εργασία της οικογενείας, της αλληλεγγύης και της συνεργασίας σχολείου, κοινωνίας και οικογενείας. Πρότεινα και ορισμένες λύσεις και πρέπει να πω ότι εις την κατά την εξέλιξη ενός ανηλίκου πρέπει να συνεργαστεί η οικογένεια με το ε, σχολείο, με τους δασκάλους και η συνεργασία γονέων και δασκάλων είναι πολύ σημαντική. Είναι σημαντική για να μπορέσει να διαμορφωθεί και ε, να εντοπιστεί αν υπάρχει κάποια κλίση προς εγκληματικές πράξεις. Είναι πολύ σημαντική δε η εξέλιξη για τους ανηλίκους, να ξέρουμε δηλαδή εγκαίρως εάν υπάρχουν υπόνοιες ε, εγκληματικότητες οποίες πρέπει να καταπολεμήσουμε. Μίλησε για το σχολείο, για την οικογένεια, αλλά παίζουν σημαντικό ρόλο και τα μέσα ενημέρωσης και ιδίως το διαδίκτυο. Αυτό που είναι βασικό είναι και ορισμένα παιχνίδια στο υπολογιστή που υποκινούν τους νέους να προβούν σε εγκληματικές πράξεις. Σε μία προηγούμενη συζήτηση μου είχε λεχθεί ότι και τα περιθωριακά άτομα είναι επιρρεπείς σε εγκληματικές πράξεις ή παραδείγματος χάρη πρόσφυγες και μετανάστες οι οποίοι βρίσκονται σε πολύ δυσχερή ε, κοινωνικο-οικονομική κατάσταση γι' αυτό και βλέπουμε στις ομάδες αυτές ότι παιδιά τα οποία μεγαλώνουν σε αυτή την ομάδα έχουν τάση προς εγκληματικότητα και γι' αυτό θεωρώ ότι πρέπει να τονίσουμε την μηδενική ανοχή από τους, ε, ε, ε, για τους ενήλικες οι οποίοι υποκινούν τους ανήλικες να διαπράξουν εγκλήματα. Ε, για να μπορέσουμε να εξασφαλίσουμε και πρόληψη ε, και επιπλέον πρέπει να τονίσουμε τα προγράμματα ε, επαναφοράς και επανακοινωνικοποιήσεως όπως επίσης και τα προγράμματα καταπολέμησης της χρήσης ναρκωτικών διότι όλες αυτές οι συμπεριφορές συμβάλλουν εις την εγκληματικότητα και πρέπει κανείς να προλάβει την ε, βία. Είναι πολύ σημαντικό να υπάρξει σωστή ε, ε, σωστή ανατροφή από την οικογένεια και θα πρέπει να υπάρχει οικογενειακός ιστός μεταξύ των παππούδων και των εγγονών γιατί η τρίτη γενιά μπορεί να επηρεάσει θετικά τους νέους. Πρέπει λοιπόν όλοι να συνεργαστούν κατά τρόπον ώστε οι γονείς να μπορέσουν να αφιερώνουν πολύ ε, χρόνο ή στην ε, ε, ανατροφή των παιδιών τους και χρειάζεται να καλυφθεί το χαμένο έδαφος για να μπορέσει να αποκαλύψει κατασταθεί ο οικογενειακός ιστός, διότι αν εργάζονται οι γονείς πρέπει συγχρόνως να έχουν τη δυνατότητα να ε, ε, εξασφαλίσουν καλή ε, περίθαλψη και εκπαίδευση των παιδιών τους. Υπάρχουν σε ορισμένες χώρες ε, ε, προσχολικά ιδρύματα τα οποία παίζουν ένα πολύ θετικό ρόλο και πρέπει να υπάρξει η οικονομική ενίσχυση ε, και προώθηση των συστημάτων που λειτουργούν ικανοποιητικά. Θα μπορούσε κανείς να πει πολλά εδώ, αλλά η συνάδελφος θέλω να ευχαριστήσω τη συνάδελφο Κορνέλησεν και την ε, κυρία Νικολάη διότι έχω προσπαθήσει να ε, λάβω υπόψη της, ε, τα σχόλιά τους. Σας ευχαριστώ για την προσοχή σας και είμαι στη διάθεσή σας για ενδεχόμενες ερωτήσεις. Σας ευχαριστούμε κυρία Ζαμπόρσκα. Κύριε Κορνέλισεν, είστε η πρώτη που ζητήσετε το λόγο. Παρακαλώ. Ευχαριστώ, κυρία Πρόεδρε. Δεν είχαμε αρκετό χρόνο για να μελετήσουμε εντελεχώς το θέμα. Φαίνεται ότι η έκθεση αυτή προχωράει με κάποιες εξάρσεις, αλλά με μεγάλα διαστήματα στο μεταξύ αυτών των εξάρσεων. Είχαμε κάποια πρόοδο σε σχέση με την προηγούμενη παραλλαγή της έκθεσης, αλλά η πρόοδος δεν είναι αρκετή, δεν είναι ικανοποιητική. Δεν είμαι πεπισμένος ότι η ισότητα των φύλων και η ε, παραβατικότητα των νέων είναι αλληλένδετες έννοιες. Παρά τις διαφορές μεταξύ ε, μεταχείρισης των αυτούργων και των θυμάτων ανάλογα με το φύλλο τους. Πάντως η έκθεση παρά είναι ευρεία, δεν επικεντρώνεται σε αυτό το σημείο και ακριβώς αυτή η διάχυση της έκθεσης με μπερδεύει κάπως. Την τελευταία φορά συζητήσαμε στη συνεδρίαση των συντονιστών τι θα κάνουμε με το έγγραφο αυτό. Είπαμε καλύτερα να το αναπέμψουμε για μια αναδιαμόρφωση προκειμένου να έχουν την ευκαιρία οι πολιτικές ομάδες να υποβάλουν τις προτάσεις τους και να το, να τροποποιήσουν. Έκανα ό,τι μπορούσα, κατέθεσα και εγώ πολλές τροπολογίες, αλλά δεν τις ε, βρίσκω και πολύ στο έγγραφο αυτό. Δεν ελήφθησαν υπόψη οι προτάσεις που έκανα. Και λυπούμε ειλικρινά για το ότι αγνοήθηκαν οι προτάσεις μου και δεν είμαι πεπισμένη ότι ως Επιτροπή Γυναικών θα πρέπει να συνεχίσουμε την ανασχόληση με την έκθεση αυτή. Ευχαριστούμε κυρία Κονέλης και κυρία Παπαδοπούλου. Ευχαριστώ. Ομολογώ ότι συμφωνώ με την προλαλή σας, ε, με την κυρία Κορνέλισον γιατί διαβάζοντας την έκθεση αποκόμισε την εντύπωση ότι έγιναν μεν κάποιες αλλαγές, αλλά λίγες. Κατάλογος των παραγόντων που επηρεάζουν την ενική παραβατικότητα, αλλά κυρίως ευθύνεται η οικογένεια, κυρίως στις οικογένειες χωρισμένων γονιών. Δηλαδή, αν ένας νέος ε, ε, προέρχεται από οικογένεια χωρισμένων, έχει μεγαλύτερη προδιάθεση στο έγκλημα, είναι πιο επιρρεπή στο έγκλημα. Δεν νομίζω ότι ισχύει κάτι τέτοιο. Έχουμε διάφορα ψηφίσματα του Συμβουλίου τη Ευρώπη και μάλιστα βλέπω μπροστά μου μία από τι συστάσει του Συμβουλίου τη Ευρώπη, τη σύσταση 2025 ε, προς ε, την Επιτροπή Υπουργών των Κρατών αναφέρεται ότι η ελληνική παραβατικότητα ε, έχει πολύμορφο και διακλαδικό χαρακτήρα και ε, εξαρτάται από πολλούς παράγοντες. Η οικογένεια, σχολείο, το περιβάλλον, η κοινωνία, όλοι αυτοί οι παράγοντες συμβάλλουν στην διαμόρφωση της συμπεριφορά του νέου. Δεν θα πρέπει να γνώμε λοιπόν από τις συστάσεις του Συμβουλίου της Ευρώπης, γιατί στην σύσταση αυτή εκδηλώνεται ιδιαίτερο ενδιαφέρον για τις ε, εθνικές μειονότητες, τις νέες γυναίκες, τις ειδικές ομάδες και τα ειδικά προγράμματα παρέμβασης και υπάρχουν πολλές συμβάσεις και καλές προτάσεις στην σύσταση του Συμβουλίου της Ευρώπης και καλό θα ήταν να ληφθούν υπόψη από την κυρία Ζαμπόσκα στην έκθεσή της. Πάντως εμείς σοσιαλιστές και δημοκράτες έχουμε την εντύπωση ότι το κοινωνικό περιεχόμενο και η επίπτωση των άλλων και πέραν του κύκλου τη οικογένεια λοιπόν θα πρέπει να ληφθούν περισσότερο υπόψη γιατί η συγκίτρια εστιάζεται υπερβολικά στο ρόλο τη οικογένεια. Ευχαριστώ πολύ, κυρία Παπαδοπούλου. Η Κυρία Τόμσον είναι η επόμενη μιλήτρια. Διάβασα και εγώ την έκθεση. Πιστεύω ότι μερικές από τις σημαντικότερες αιτίε ε, για την ελληνική παραβατικότητα δεν περιλαμβάνονται σε αυτό το εγγραφό. Αυτό που είναι περίεργο είναι ότι σχετίζεται τους γονείς, τους εργαζόμενους γονείς με το έγκλημα στους νέους ανθρώπους. Όλα τα στατιστικά στοιχεία δείχνουν ότι οι άνεργοι μετανάστες γονείς ε, παραμένουν τα παιδιά που παραμένουν παιδιά, με τα παιδιά όλη τη μέρα έχουν τη μεγαλύτερη παραβατικότητα μεταξύ των νέων. Επισκέφθηκα ένα μέρος της Σλοβακία όπου 90% των Ρωμά ήταν σπίτι όλη μέρα. Τα παιδιά δεν πήγαιναν στο σχολείο, ήταν εγκληματίε και υπήρχαν πολλά προβλήματα. Δεν καταλαβαίνω λοιπόν ποια είναι η σχέση μεταξύ εργαζομένων γονέων και νέων που ε, έχουν υψηλή παραβατικότητα. Βλέπουμε επίσης περίπτωση των ε, μονογονεϊκών οικογενειών με τη μητέρα μόνο όταν δεν εργάζονται, είναι σπίτι όλη μέρα, δεν ανήκουν στην αγορά εργασίας τότε έχουν προβλήματα. Όταν δουλεύουν, κερδίζουν χρήματα, είναι χαρούμενες με άλλους ενήλικες όλη μέρα, δεν δημιουργούν παιδιά που ε, καταφεύγουν στο έγκλημα. Δεν καταλαβαίνω λοιπόν ποια είναι η λογική του να οι άνθρωποι να παραμένουν μακριά από την αγορά εργασία και να φροντίζουν τα παιδιά. Είναι σημαντικό να έχουμε Καλού θεσμού Βρήκαμε μια οικογένεια στη Δανία με 10 παιδιά, ήταν κατά των αμβλώσεων και σήμερα είναι σπίτι όλη μέρα και δυστυχώς τώρα πολύ αργά οι κοινωνικές αρχές τους βρήκαν και τους έβγαλαν από αυτό το σπίτι. Ταξιδεύοντας στην Ευρώπη βλέπω φρικτές συνθήκες για τα παιδιά. Πιστεύω ότι είναι πρόβλημα που δεν παίρνουμε αρκετά παιδιά από το σπίτι τους σε καλούς θεσμούς επειδή πολλοί γονείς δεν είναι ικανοί να είναι καλοί γονείς. Εάν είναι ικανοί μόνο κατά το ίμιση, τότε οι δημοσίοι θεσμοί, τα νηπιαγωγεία, τα σχολεία, οι οργανώσεις για τους νέους μπορούν να αντισταθμίσουν όσα δεν μπόρεσαν να παρέχουν οι γονείς. Χρειαζόμαστε λοιπόν αυτήν όλη την προοπτική πώς θα σώσουμε παιδιά από δυσλειτουργικά σπίτια. Το χειρότερο πράγμα για ένα παιδί είναι με γονεί δυσλειτουργικού είναι το να παραμένει στο σπίτι αντί να βρίσκεται σε ένα νηπιαγωγείο το οποίο του παρέχει κίνητρα. Ευχαριστώ κυρία Τόμσον. Η κυρία Νίκολαη είναι η επόμενη ομιλήτρια. Δυστυχώς ε, αυτή είναι έκδοση. Δεν είναι αυτό που περίμενα. είναι λίγο πιο μπερδεμένη και λίγο ασαφής όσον αφορά το θέμα της. Το θέμα είναι δύσκολο σε κάποιο βαθμό. Είναι δύσκολο να το μελετήσει κανείς, να δημιουργήσει σχέση αιτίας και αποτελέσματος μεταξύ της ισότητας των ευκαιριών και της παραβατικότητας των νέων. Θα προσπαθήσω όμως να είμαι θετική. Επειδή έχω υποβάλει ήδη πολλές τροπολογίες προσπαθώντας να βελτιώσω την ποιότητα της εργασίας. Αν θα ήταν δυνατό με την προθεσμία, αν μπορούσαμε να κάνουμε κάτι με την προθεσμία υποβολής των τροπολογιών, θα μπορούσαμε να καταλήξουμε σε ένα κείμενο καλής ποιότητας, αλλά έτσι όπως έχουν τα πράγματα με όλα αυτά τα ασαφή ερωτήματα όσον αφορά τη δυνατότητα να ξεκινήσουμε μια, ένα προβληματισμό για την πολιτική ίσων ευκαιριών. Έχουν ξεκινήσει αυτοί οι προβληματισμοί εδώ και πολύ καιρό. Αυτή τη στιγμή αναπτύσσουμε το θέμα και υπάρχουν και άλλα σχετικά ερωτήματα. Εάν είχαμε αυτή τη στιγμή την ευκαιρία να υποβάλουμε τροπολογίες, ε, παραδείγματο χάρη το Σεπτέμβριο, επειδή δυστυχώ την επόμενη εβδομάδα είναι μια πράσινη εβδομάδα και τελειώνει η περίοδος, ε, θα μπορούσαμε να βελτιώσουμε την έκθεση από αυτή την άποψη. Ευχαριστώ κυρία Νικολάη. Η επόμενη μιλήτρια είναι η αντιπρόσωπος της Επιτροπής, η κυρία Μυρίνα. Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ για αυτή την ενδιαφέρουσα συζήτηση και για το σχέδιο γνωμοδότησης. Άκουσα όλους σας με πολύ προσοχή και θα επανέλθω με περαιτέρω σχόλια στην επόμενη συνάντησή μας. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ κυρία Μπάουερ, ζήτησε το λόγο. Ευχαριστώ πολύ. Ένα σύντομο σχόλιο για τη συζήτηση και όσον αφορά την έκθεση. Ενίοτε αντιμετωπίζουμε ζητήματα τα οποία βρίσκονται στα όρια αρμοδιοτήτων και ευθύνης ε, διαφορετικών επιτροπών. Ίσως αν τούτου είδου η έκθεση να ήταν καταλληλότερη για την Επιτροπή ΛΥΜΠΕ, για την Επιτροπή Πολιτισμού. Δεν ξέρω, ίσως και για κάποια άλλη Επιτροπή. Αναμφίβολα. Η παράλληλη ύπαρξη της επαγγελματικής και της ιδιωτικής ζωής ε, επηρεάζει αυτό το ζήτημα. Μερικές φορές είναι δύσκολο να συλλάβουμε ποια είναι η σωστή ισορροπία. Ωστόσο, οι οικογενειακές ε, υποχρεώσεις ε, αναμφίβολα. Συμφωνώ απόλυτα. Έχουμε οικογένειες που πουλάνε παιδιά, έχουμε οικογένειες που είναι δυσλειτουργικές. Υπάρχουν ε, πολύ, πολλές και διαφορετικές πραγματικότητες όσον αφορά τις οικογένειες. Έχω την αίσθηση ότι είναι πολύ δύσκολο να βρει κανεί ε, το επίπεδο, το απαιτούμενο επίπεδο όπου μπορούμε να έχουμε μια ολοκληρωμένη άποψη επειδή η πραγματικότητα είναι τόσο κατακαιρματισμένη, τόσο διαφοροποιημένη. Έχω ωστόσο την αίσθηση ότι θα πρέπει να προσπαθήσουμε να διαμορφώσουμε μια δική μας ιδιαίτερη συμβολή προς την επίλυση και την αντιμετώπιση αυτού του ζητήματος. Σας ευχαριστούμε κυρία Μπάουερ. Κυρία Ζαβόρσκα, έχετε το λόγο. Ευχαριστώ θα κάνω ορισμένα σχόλια. Δεν συμφωνώ απολύτως. Δεν θα συμφωνήσω με τους συναδέλφους που λέγουν ότι εγώ ε, επιμένω υπερβολικά στην ε, οικογένεια διότι ε, θεωρώ ότι όντως ε, επηρεάζουν ε, την εξέλιξη των νέων, ιδίως όσον αφορά την εγκληματικότητα. Πρέπει κανείς να συνδυάζει την οικογενειακή ζωή με την επαγγελματική πορεία και ο συνδυασμός αυτός ε, είναι αναγκαίο γιατί αν τον επιτύχουμε θα μειώσουμε και θα επηρεάσουμε θετικά την, την εγκληματικότητα των νέων. Υπάρχουν πολλές πληροφορίες που αποδεικνύουν ότι ο χρόνος που διαθέτουν οι γονείς στα παιδιά επηρεάζει την περαιτέρω πορεία του στη ζωή. Δεν είναι ο μοναδικός παράγων ο οποίος μπορεί να προλάβει την εγκληματικότητα. Δεν είναι δηλαδή μία σαφής ξεκάθαρη κατάσταση άσπρο ή μαύρο, αλλά όσο περισσότερο χρόνο περνάει ο γονιός χρόνο με τα παιδιά τόσο περισσότερο τα επηρεάζει χωρίς όμως αυτό να σημαίνει ότι δεν πρέπει να μας ενδιαφέρει ο συνδυασμός επαγγελματικής και οικογενειακής ζωής. Η πιο εκτενής ε, παράγραφος ε, της εκθέσεώς μου είναι αυτή όπου εξετάζουμε τις προϋποθέσεις που μπορούν να οδηγήσουν ε, σε εγκληματικότητα. Διότι και ε, και οι ναρκωμανείς ε, οδηγούνται στην ε, εγκληματικότητα. Μία ομιλήτρια αναφέρθηκε στις οικογένειες Ρωμά, αλλά οι οικογένειες αυτές είναι διαταραγμένες, μπορεί να ζουν κάτω από την ίδια στήχη, στέγη, αλλά είναι οικογένειες όπου πολλές φορές οι γονείς δεν εργάζονται, τα παιδιά δεν πηγαίνουν σχολείο και υποκινούνται να εγκληματίσουν. Πρέπει να μιλάμε για μία εύρυθμα λειτουργούσα οικογένεια ε, ε, εκεί να δούμε ε, πώς το παιδί μπορεί να οδηγηθεί στην εγκληματικότητα και υπάρχει το θέμα της ε, φτώχειας, της περιθωροποιήσεως, της ε, εκπαιδεύσεως, της παιδείας ε, για τα παιδιά. Προσπάθησα να, να απαριθμίσω όλους τους παράγοντες ε, δεν ε, τους επινόησα εγώ, αλλά βασίστηκα στους ορισμούς οι οποίοι υπάρχουν και πρόκειται για τους ορισμούς ε, που βρίσκουμε σε επίσημα έγγραφα. Βέβαια προφανώς ε, θα μπορούσε να προσθέσει κανείς διάφορα σε αυτή την έκθεση διότι το θέμα είναι πολύ ευρύ όπως το είπε και η κυρία Μπάουερ θα μπορούσαν ε, εδώ να επιληφθούν ε, και να είναι αρμόδιες διάφορες ε, επιτροπές αλλά δεν είναι η πρώτη φορά. Πολλές φορές ε, είχαμε ε, διάφορες επιτροπές ε, που συνεργάστηκαν ή που απέριπταν τις τροπολογίες διότι θεώρησαν ότι ήταν άλλης επιτροπής αρμοδιότητας η έκθεση αυτή. Ευχαριστώ για όλα τα σχόλια, αλλά ενδεχομένως ορισμένα δεν συνάδουν με τις προθέσεις μου. Προσβλέπω στις τροπολογίες σας, τις οποίες θα κοιτάξω να ενσωματώσω, αλλά είχα την εντύπωση ότι πολλά σχόλια υποκινούνται από πολιτικές σκοπιμότητες και γι' αυτό το λόγο δεν μπορούμε να καταλήξουμε σε μία ενιαία λύση. Οπότε θα παρακαλέσω την Πρόεδρο να μας πει τι χρονοδιάγραμμα προβλέπει για αυτή την έκθεση ε, και αύριο θα μέχρι αύριο θα αποφασίσω αν θα συνεχίσω αυτή την έκθεση ή όχι. Σας ευχαριστούμε κυρία Ζάμπορσκα. Όπως είχαμε προβλέψει και στην αρχή, η διορία για την κατάθεση τροπολογιών λύγει στις 15 Ιουλίου το μεσημέρι. Όντως ο χρόνος ε, είναι σύντομος. Αυτή η προθεσμία είναι αρκετά σύντομη, γι' αυτό σπεύστε να καταθέσετε τροπολογίες. Θα ήθελα να ζητήσω και τη γνώμη των ε, σχεδόν εισηγητών και των υπολείπων μελών. Πιστεύετε μήπως ότι χρειάζεται παράταση της προθεσμίας για την κατάσταση τροπολογιών. Σε τέτοια περίπτωση όμως δεν θα προλάβουμε να είμαστε έτοιμοι για το Σεπτέμβριο. Καταρχήν εσείς κυρία Ζαμπόρσκα που είστε συγκεκριά. Τι γνώμη έχετε για την, για την προθεσμία. Κύριε Πρόεδρε ευχαριστώ. Εάν ε, με τα κυλήσει η ψηφοφορία μέχρι μέση Σεπτεμβρίου ε, ενδέχεται να μεταφέρουμε και την ε, προθεσμία ε, για την υποβολή τροπολογιών στην πρώτη εβδομάδα του Σεπτεμβρίου. Πιστεύετε ότι είναι εφικτό αυτό? Om 15 Καλώς θα το εξετάσουμε. Αν πούμε 15 Σεπτεμβρίου, για την ψηφοφορία, τότε μπορούμε να παρατείνουμε μέχρι τις 29 Αυγούστου την διορία για τις τροπολογίες. Συμφωνείτε? Ποια είναι η γνώμη και των υπόλοιπων συναδέλφων. Περιμένω τις αντιδράσεις σας. Έχω υπόψη ότι το θέμα αυτό βρίσκεται επιτάπητος εδώ και πάρα πολύ καιρό. Μπορούμε να ψηφίσουμε στις 15 Σεπτεμβρίου στην Επιτροπή, οπότε η διορία για τις τροπολογίες να λύγει στις 29 Αυγούστου. Συμφωνείτε? Θεωρείτε ότι είναι σκόπιμη η παράταση της προθεσμίας για την υποβολή τροπολογιών μέχρι τις 29 Αυγούστου, κύριε Κορνέλισεν. Κυρία Πρόεδρε, αρχικά είχαμε προβλέψει να ψηφίσουμε στις 15 Σεπτεμβρίου, ούτως ή άλλως δεν άλλαξε τίποτα δηλαδή. Οπότε, αν η διορία για τις τροπολογίες λήξει στις 29 Αυγούστου, αναβολή δεν προβλέπεται για την ψηφοφορία, γιατί είναι σημαντικό να προβλέψουμε και το χρόνο για, τα, για τις εκθέσεις πρωτοβουλίας. Γιατί έχουμε πολλές ιδέες και εκεί μας πιέζει ο χρόνος, να μην χάσουμε την ευκαιρία να υποβάλουμε και τέτοιες εκθέσεις πρωτοβουλίας. Ja, jag ska försöka er. Jag blev också lite fundersam. Μάλιστα, πρέπει να παραδεχτώ ότι χρειάστηκε να το σκεφτώ αυτό 29 Αυγούστου και παρόλα αυτά μπορούμε πάλι να ψηφίσουμε στις 15 Σεπτεμβρίου. Δεν είμαι σίγουρη πως αυτό θα μπορούσε να λειτουργήσει επειδή είχαμε την προτινόμενη προθεσμία της 15 Ιουλίου, το προτείναμε διότι αναμέναμε πολλές τροπολογίες. Γι' αυτό θεωρήσαμε ότι χρειαζόμασταν αρκετό χρόνο πριν το θέσουμε σε ψηφοφορία το Σεπτέμβριο. Αυτό είχαμε σκεφτεί αρχικά. Αν το επιθυμείτε μπορούμε να παρατείνουμε μέχρι τις 29 Αυγούστου την προθεσμία για την υποβολή τροπολογιών έχοντας υπόψη μας ότι αν λάβουμε πολλές αλλά πραγματικά πολλές τροπολογίες τότε θα χρειαστεί να αναβάλουμε και την ψηφοφορία τον Οκτώβριο. Στόχος μας είναι να το κάνουμε έγκαιρα 29 Αυγούστου για τις τροπολογίες προθεσμία και να το ψηφίσουμε για τις 15 Σεπτεμβρίου. Συμφωνούμε με αυτό το χρονοδιάγραμμα. Η κυρία Τόμσεν. Δεν ακούγεται το μικρόφωνο. Ε, πιστεύω ότι καλό θα ήταν ε, να αναβάλουμε την υποβολή τροπολογιών μέχρι τις 29 Αυγούστου. Κυρία Τόμσεν, ε, πολύ καλά. Η συγγήτρια φαίνεται να συμφωνεί με την κυρία Τόμσεν και πολλά μέλη επίσης, αν κρίνω από τα νεύματά τους, 29 Αυγούστου 5 μετά μεσημβρίας, προθεσμία για την υποβολή τροπολογιών, πολύ καλά. Ευχαριστώ για την ενδιαφέρουσα συζήτηση και για τις επικοδομητικές προτάσεις σας για το πώς πρέπει να προχωρήσουμε στη συνέχεια. Έχουμε ακόμα ένα στοιχείο στην ε, ημερήσια διάταξη. Ας προσπαθήσουμε να το κάνουμε και αυτό σήμερα. Η κυρία Σαπόσκα, πάλι είναι το σχέδιο γνωμοδότησης που θέλουμε να υποβάλουμε στην Επιτροπή Απασχόλησης και Κοινωνικών Υποθέσεων αφορά την Ευρωπαϊκή Πλατφόρμα κατά της ένδυας και, κοινωνική, και του κοινωνικού αποκλεισμού. Θα ήθελα να σας υπενθυμίσω ότι αυτή η Ευρωπαϊκή Πλατφόρμα είναι μία από τις εμβληματικέ πρωτοβουλίες που έχει υποβάλει η Κομισιόν στο πλαίσιο της στρατηγικής Ευρω... 2020 ε, ε, ας μας, δώσει, ας μας μιλήσει η συγκήτρια για την γνωμοδότηση. Κυρία Ζαμπόσκα. Ευχαριστώ κυρία Πρόεδρε. Όπως και εσείς είπατε, η πλατφόρμα αυτή ε, για την ε, καταπολέμηση ε, της φτώχειας και του κοινωνικού αποκλεισμού είναι ένα από τα πολλά θέματα που εξετάζει η Επιτροπή μας. Πρέπει όμως να σας πω από την αρχή ότι από όταν εγώ ε, συμμετέχω στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και είμαι εδώ ήδη 7 χρόνια και πρέπει να σας πω ότι δεν ξέρω τι, ε, πόσες γνωμοδοτήσεις έχουμε κάνει σχετικά με την φτώχεια και την καταπολέμησή της στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Πριν λίγο καιρό ήταν το Ευρωπαϊκό έτος κατά της φτώχειας και πρέπει να σας πω από την ε, ευθύ ε, εξ αρχή ότι η κατάσταση είναι τέτοια ώστε ε, έχουμε συνέχεια νέα έγγραφα τα οποία υιοθετούμε αλλά η κατάσταση δεν βελτιώνεται. Δηλαδή δεν είναι αρκετά αποτελεσματική η ε, πρόοδος. Προσπάθησα στα πλαίσια αυτά να ζητήσω από την Ευρωπαϊκή Ένωση και να την καλέσω να κάνει μία απογραφή της κατάστασης ε, της φτώχειας. Χρειαζόμαστε αξιόπιστα στατιστικά στοιχεία και νομίζω ότι τα στοιχεία τα οποία έχουν δημοσιευθεί και ε, που προβαίνουν σε διάφορους ορισμούς της στόχιας δεν συμβάλλουν ε, στην βελτίωση της καταστάσεως. Θα έπρεπε να υπάρχουν πιο συγκεκριμένα ε, κείμενα και ερευνές να διαχωρίσουμε την φτώχεια στις άντρες από αυτήν στις γυναίκες να υπάρξει ένας ορισμός ε, του, τι εννοούμε ε, ε, με τους όρους εμπορεύματα και υπηρεσίες γιατί στη φτώχεια δεν έχουμε αρκετούς καλούς ορισμούς για να προβούμε σε μια σωστή οριοθέτηση. Ένα άλλο θέμα το οποίο με απασχολεί είναι η οικονομική και κοινωνική κατάσταση των οικογενειών που καταλήγει στο ότι τα παιδιά ε, οδεύουν προς ε, κοινωνικές ε, κοινωνικές ε, εγκαταστάσεις ε, που είναι η βάρος της περαιτέρω εξελίξεώς τους. Θα πρέπει τα παιδιά να μπορούν να μείνουν στον πυρήνα της οικογένειας ή τουλάχιστον να μπορέσουν να αναλυφθούν από μία εναλλακτική οικογένεια όσο καιρό διαρκεί η κατάσταση της ένδυας στην οικογένειά τους. Πιστεύω ότι σήμερα η φτώχεια ε, θα πρέπει να αποτελέσει προτεραιότητα της Ευρωπαϊκής Επιτροπής κατά τρόπον ώστε να υπάρξει ένα ειδικό τμήμα για την φτώχεια και ε, ο πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Ένωσης θα έπρεπε επίσης να γνωμοδοτήσει επί της φτώχειας όπου θα αναφέρει την κατάσταση των ανδρών και των γυναικών. Ε, και τέλος θα ήθελα να πω ότι η ε, οργάνωση θεμελιωδών δικαιωμάτων θεωρεί ότι η ακραία ε, ένδια αποτελεί μία παραβίωση των θεμελιωδών δικαιωμάτων. Παρακαλώ λοιπόν τον οργανισμό αυτόν ο οποίος ε, ε, να ασχοληθεί με αυτά τα θέματα εφόσον ο οργανισμός αυτός είναι ένα από τα θεσμικά όργανα της Ευρωπαϊκής Ενώσεως. Ευχαριστώ κυρία Ζαμπόρσκα. Είναι η κυρία Μπλινκεβιτσούτε. Ευχαριστώ κυρία Πρόεδρε. Θα ήθελα να ευχαριστήσω και εγώ θερμά την εισηγήτρια, την κυρία Ζάμπορσκα, για την έκθεσή της και συμφωνώ απόλυτα μαζί της ότι μπορούμε να εκπονούμε όσε εκθέσει θέλουμε και γνωμοδοτήσει, αλλά αυτό δεν οδηγεί σε πραγματική μείωση τη φτώχεια τη χώρα. Βέβαια, το φαινόμενο αυτό συνδέεται και με την παγκόσμια οικονομική και χρηματοπιστωτική κρίση. Αυτό όμω δεν σημαίνει κατά ανάγκη ότι θα πρέπει να σταυρώσουμε τα χέρια και να παραιτηθούμε από την προσπάθεια καταπολέμησης ε, της φτώχειας και εδώ στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Η Επιτροπή μας είναι η Επιτροπή των Δικαιωμάτων των Γυναικών και της Ισότητα των Ευκαιριών. Δεν πρέπει λοιπόν να ξεχνάμε ότι οι γυναίκες είναι αυτές που πιο συχνά πέφτουν στην παγίδα της φτώχειας. Και αυτό θα πρέπει να το τονίσουμε στην έκθεση. Συμφωνώ ότι χρειαζόμαστε σαφή και συγκεκριμένα στοιχεία για τις διαστάσεις που έχει το φαινόμενο της φτώχειας. Και αυτά τα συγκεκριμένα στοιχεία θα αποτελέσουν τη βάση για σωστές πολιτικές αποφάσεις. Επίσης πρέπει να γίνει μία ε, διάκριση των δεδομένων ανάλογα με το φύλλο και την ηλικιακή ομάδα. Για παράδειγμα, θέλουμε στοιχεία για ηλικιωμένε γυναίκες και πώς αυτές ε, πλήττονται από τη φτώχεια. Είναι πολύ, τέτοια, είναι πολύ χρήσιμα τέτοια στοιχεία ανά κατηγορία. Επίσης ε, θα πρέπει να υποβάλουμε συγκεκριμένες προτάσεις, για παράδειγμα μέτρα που θα ενισχύσουν την απασχόληση και την ε, εκπαίδευση των γυναικών ή θα εξομοιώσουν τις μισθολογικές διαφορές μεταξύ ανδρών και γυναικών. Τέτοιου είδους ζητήματα θα πρέπει να περιλάβουμε στην έκθεση. Θα ήθελα επίσης να σας επιστήσω την προσοχή στο γεγονός ότι πολύ συχνά οι μονογονεϊκές οικογένειες είναι οι πιο ευάλωτες στη φτώχεια. Ας μην το ξεχνούμε και αυτό και να το τονίσουμε, να δούμε και να απευθύνουμε έκκληση στα κράτη-μέλη να στηρίξουν τις μονογονεϊκές οικογένειες για να αποφύγουν το φάσμα της φτώχειας. Ένα άλλο θέμα αφορά την οδηγία για το ελάχιστο εισόδημα. Αν δεν καταλήξουμε σε συμφωνία ως προς το ελάχιστο εισόδημα, θα αποτύχουμε στην προσπάθειά μας να πατάξουμε τη φτώχεια. Θα πρέπει πρώτα να διεκπαιρεώσουμε ε, τις εργασίες για την οδηγία για το ελάχιστο εισόδημα. Αυτό θα είναι σημαντικό εργαλείο για την καταπολέμηση της φτώχειας. Συμφωνώ απόλυτα με την εισηγήτρια ότι η Επιτροπή θα πρέπει να συγκροτήσει μία μονάδα που θα έχει αποκλειστικό στόχο την καταπολέμηση της φτώχειας. αλλά διαρωτώ με, δεν έχει ήδη αρκετέ μονάδε και διευθύνσει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Χρειάζεται μια επιτούτου μονάδα. Ε, ε, Χρειαζόμαστε και συγκεκριμένα μέτρα σε τοπικό και περιφερειακό επίπεδο, ιδιαίτερα στην Ήπεθρο, στις αγροτικές ζώνες και να επικεντρωθούμε και στις ζώνες αυτές, στα προβλήματα των ηλικιωμένων, στου αναπήρους, στις γυναίκες αλλά και τους άντρες και στο πλαίσιο αυτό θα ήθελα να αναφερθώ στην οδηγία για τις κοινοφελείς υπηρεσίες και την πρόσβαση στις υπηρεσίες αυτές. Γιατί η εξασφάλιση πρόσβαση στις κοινοφελείς υπηρεσίες είναι επίσης εργαλείο για την καταπολέμηση της φτώχειας. Εστερνίζομαι τη γνώμη σας για, για τον οργανισμό θεμελιωδών δικαιωμάτων ή βασικών δικαιωμάτων, αλλά ένας τέτοιος οργανισμός θα πρέπει να έχει στερή συνεργασία με το Ινστιτούτο για την Ισότητα των Φύλων. Έτσι θα διευκολύνουμε και την σύναψη συμβαστικών λύσεων. Πιστεύω ότι θα καταλήξουμε σε μια πολύ καλή γνωμοδότηση. Ευχαριστώ πολύ κύριε Τόμσεν. Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστούμε για την γνωμοδότηση η οποία πιστεύω είναι εξαιρετική και συμφωνώ επίσης ε, με τα στατιστικά στοιχεία είναι πολύ σημαντικό και για όσα είπε η κυρία Μπλινκοβίτς για ε, τις αρρωγές να ψάξουμε να βρούμε πού είναι οι φτωχότεροι άνθρωποι αίσθησή μου είναι ότι σήμερα στην Ευρώπη παρατηρούμε μια νέα τάση, νέες κοπέλες που αποκτούν πολλά παιδιά. Έχω δει ντοκιμαντέρ στην τηλεόραση από το Ηνωμένο Βασίλειο, από τη δική μου χώρο, όπου 24χρονες ανήπαντρες μητέρες έχουν 5 παιδιά και αναρωτιέμαι τι είδους φαινόμενο είναι αυτό. Δεν συνέβαινε στην ίδια έκταση πριν από 20 χρόνια. Και έτσι παράγεται ένδια με όλα αυτά τα παιδιά σε νέα ηλικία. Αυτή η γυναίκα δεν έχει εκπαίδευση. Έχει να κάνει όλο αυτό με την ε, έλλειψη της σεξουαλικής εκπαίδευσης στα σχολεία. Όπως συνέβαινε βέβαια και σε παλιότερες εποχές ε, ε, ακούγεται λίγο αντιδραστικό, αλλά αυτός ε, είναι και ο λόγος που κάποιες νέες γυναίκες έχουν πολλά παιδιά. Είναι παράγον που οδηγεί στην ένδυα. Δεν θα πρέπει να αποφύγουμε την εξαναγκασμένη, τον εξαναγκασμένο εκτοπισμό παιδιών από τις ε, κακές οικογένειες. Δεν συμφωνώ με αυτό. πιστεύω ότι υπάρχει ένα σημαντικό ζήτημα στο σημείο 6 όπου συζητάτε με την πραγματική πρόσβαση των φτωχότερων στα θεμελιώδη δικαιώματα. δεν μελετά, έχουμε μελετήσει επαρκώς την πρόσβαση αυτή στα θεμελιώδη δικαιώματα, διότι οι φτωχοί άνθρωποι πολύ συχνά σε όλη την Ευρώπη δεν μπορούν να έχουν πρόσβαση σε αυτά τα δικαιώματα. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ κύριε Τόμσεν. Κυρία Παπανόβα, ευχαριστώ κυρία Ζαμπόσκα για την έκθεση και ελπίζω ότι αυτή θα έχει καλύτερη μοίρα. Ε, κοιτώντας την πιστεύω ότι θα καταφέρουμε να συμφωνήσουμε. Επικριτώ τον τρόπο που αντιμετωπίζετε τι διαφορέ τη ένδυα και ειδικότερα όταν μιλάτε για την πρόσβαση στην εργασία, την κοινωνική ασφάλιση, τι ουσιώδει υπηρεσίε αλλά φυσικά και τα ζητήματα υγείας είναι πολύ σημαντικά, ειδικότερα όταν μιλάμε για άτομα με αναπηρίες, χρόνιες ασθένειες. Η εκπαίδευση επίσης ε, αποτελεί, μπορεί να γίνει ένα σημαντικό εμπόδιο και να συμβάλλει σημαντικά στη λύση. μπορούμε να αντιμετωπίσουμε το ζήτημα από δύο πτυχές. Το, η μία είναι η πρόληψη της φτώχειας και η δεύτερη είναι η, ο προσδιορισμός του φαύλου κύκλου του όπου παραμένει κάποιος φτωχός και το δεύτερο κομμάτι είναι το πώς βγάζουμε τους ανθρώπους από αυτή την ένδια. Θα έλεγα ότι φυσικά αυτά που αναφέρεται για τις οικογένειες έχουν σημαντικές επιπτώσεις. Πιθανώ δίνοντα το παράδειγμα της προηγούμενη έκθεσης θα μπορούσαμε και πάλι να αποφύγουμε να τονίσουμε τόσο πολύ τι οικογένειε, διότι οι οικογένειες υπάρχουν σε διαφορετικές μορφές. Έχετε απόλυτο δίκιο, υπάρχουν πιο συντηρητικέ και θρήσκε οικογένειες και πιο νέου τύπου οικογένειε, ε, μονογονέκες. Ε, ε, ε, καμιά φορά δεν είναι, είναι κανικογένειες, είναι μόνο ένα άτομο ε, που εκτίθενται σε τεράστια φτώχεια. Ολόκληρη η κοινωνία και η οικονομική ανάπτυξη συμβάλλουν σε αυτό το φαινόμενο. Το πρόβλημα είναι δύσκολο να αναλυθεί και να συγκριθεί και να γίνουν συγκρίσεις ε, μεταξύ όλων αυτών των παραγόντων. Θα έλεγα ότι η σωστή ανάλυση είναι απολύτως ε, ζωτική σημασίας. Για αυτό το λόγο από την άποψη της επίπτωση στην οικονομική ανάπτυξη και την κοινωνική ανάπτυξη των οικογενειών. Αυτό ίσως είναι κάτι που θα ε, περάσει. Θα συνέστηνα, ωστόσο, να μην εξετάσουμε γενικότερα μόνο την οικογένεια ως πηγή της ένδυας ή ως πηγή αποφυγής της ένδυας. Θα πρέπει να ψάξουμε πιο βαθιά στους οικονομικούς παράγοντες. Γενικά όμως, σε γενικές γραμμές πιστεύω ότι αυτή η εκθέση θα είναι επιτυχής. Ευχαριστώ. Ε, Ευχαριστώ κύριε Παύλο. και πριν δώσω το λόγο ξανά στην κυρία Ζαμπόρσκα θα ήθελα να εκμεταλλευτώ την ευκαιρία για να κάνω και εγώ ίδια μερικά σχόλια. Άκουσα προσεκτικά τη συζήτηση εδώ στην αίθουσα. Θα ήθελα να ευχαριστήσω την κυρία Ζαμπόρσκα πρώτα απ' όλα και από τα σχόλια ε, και των υπόλοιπων συναδέλφων έχω την αίσθηση ότι αυτό το στοιχείο θα γίνει μια καλή γνωμοδότηση στην οποία θα μπορέσουμε να συμφωνήσουμε. Επίσης ε, συμφωνώ με όσους ε, λέγουν ότι συζητάμε πολύ συχνά για τη φτώχεια αλλά είναι πολύ δύσκολο να επιτύχουμε κάποια απτή αλλαγή ακούγοντας ε, στη συζήτηση μου ήρθε και μια άλλη σκέψη. Βλέπουμε να αυξάνεται η φτώχεια σε πολλά κράτη-μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης και παράλληλα παρατηρούμε ότι ορισμένοι άνθρωποι γίνονται περισσότεροι από ποτέ σε άλλες ομάδες της κοινωνίας. Συνεπώς έχουμε αύξηση και της φτώχειας και του πλούτου. Συνεπώς όταν μιλάμε για φτώχεια θα ήταν... Πρέπει να έχουμε υπόψη μας και αυτή την εξέλιξη με άλλα λόγια. Το χάσμα γίνεται όλο και πιο μεγάλο Υπάρχουν πολλές διαφορές όσον αφορά την πρόσβαση στις κοινωνικές υπηρεσίες και εκεί συμβαίνει το ίδιο. Οι κοινωνικές υπηρεσίες ε, είναι θεμελιώδου σημασία, ειδικότερα για τις ευάλωτες ομάδες, για τα άτομα με προβλήματα κινητικότητας, ηλικιωμένου, ασθενείς. Γι' αυτό το λόγο πιστεύω ότι θα πρέπει να συζητήσουμε και αυτό το ζήτημα, πώς μπορούμε να το χρηματοδοτήσουμε, τις κοινωνικές υπηρεσίες και να διασφαλίσουμε αυτές οι υπηρεσίες να είναι προσπελάσιμες από όσους τις χρειαζόνται περισσότερο. Επιπλέον, ήθελα να μοιραστώ κάτι άλλο μαζί σας. Στη χώρα μου, στη Σουηδία, συζητάμε σχετικά με την παιδική ένδια, η οποία αυξάνεται στη Σουηδία αυτή την εποχή. Είναι σημαντική η συζήτηση για μας. Μπορούμε να συζητήσουμε για φτώχεια σε μια πλούσια χώρα όπως η Σουηδία, σε μια χώρα ε, Κοινωνική πρόνοιας όπως είναι η Σουηδία. Μιλάμε για αυτό για τα παιδιά. Τι συμβαίνει τότε με τα παιδιά στις υπόλοιπε χώρες, στι ε, χώρε του τρίτου κόσμου. Αυτή η συζήτηση, ωστόσο, λαμβάνει χώρα αυτή τη στιγμή στη χώρα μου και θα πρέπει να το θυμόμαστε αυτό. Υπάρχουν κράτη-μέλη εντό της Ευρωπαϊκή Ένωση, που είναι σύμβολα του κοινωνικού κράτους και παρόλα αυτά βλέπουν να έχουν στις χώρες τους ε, παιδική φτώχεια. Τα παιδιά μεγαλώνουν σε πολύ διαφορετικές ε, ε, συνθήκες. Δεν έχουν την ευκαιρία να συμμετέχουν στην κοινωνία όπως θα έπρεπε. Είμαι βέβαιη ότι όλοι θέλουμε τα παιδιά να έχουν αυτό το δικαίωμα, όλα τα παιδιά. Ευχαριστώ και πάλι την κυρία Ζαμπόσκα, ευχαριστώ για την γνωμοδότησή σας. Είμαι πεπισμένη ότι μαζί θα μπορέσουμε να συγκεντρώσουμε την πλειοψηφία που χρειάζεται για την γνωμοδότησή σας. Δεν ξέρω αν υπάρχει κάποιος εδώ από την Κομισιόν για αυτό το θέμα. Δεν βλέπω να είναι κανείς. Έτσι δίνω το λόγο στην κυρία Ζαμπόσκα ώστε να μας δώσει τις τελικές της παρατηρήσεις όσον αφορά την γνωμοδότηση. Κυρία Ζαμπόσκα. Ευχαριστώ κυρία Πρόεδρε. Θα ήθελα να ευχαριστήσω για όλες τις παρατηρήσεις και η οπτική γωνία από την οποία εξετάζουμε ε, ε, την φτώχεια διαφέρει αναλόγως της τοποθέτησης. Ε, υπάρχουν οι ομάδες οι οποίες είναι πιο ευάλωτες από τις άλλες, αλλά όταν ζήτησα στατιστικά στοιχεία ανταλήφθηκα ότι δεν ήταν δυνατόν οι στατιστικές να περιλάβουν όλα αυτά τα στοιχεία και ενδεχομένως εάν ε, ζητήσουμε πάρα πολλά πράγματα από την Ευρωπαϊκή Ένωση τότε δεν πρόκειται ε, η Ευρωπαϊκή Ένωση να καταρτήσει καμία στρατηγική. Δηλαδή αυτό που θέλω τουλάχιστον είναι να υπάρχει μία κατανομή των στατιστικών μεταξύ ανδρών και γυναικών στην Επιτροπή μας ε, ψηφίσαμε και πάντοτε εγώ ήμουνα υπέρ του κατωτάτου μισθού. Πρέπει να υπάρχει ένας κατώτατος μισθός, ίσως όχι όπως το γαλλικό ΣΜΙΚ, αλλά πρέπει να υπάρχει ένας καθορισμένος, ένα καθορισμένο επίπεδο κάτω από το οποίο δεν πρέπει να πέφτει η αμοιβή της εργασίας. Ξέρω όμως ότι αυτό είναι δύσκολο και το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ενδεχομένως δεν θα συμφωνήσει στο θέμα αυτό, δηλαδή δεν είναι δυνατόν το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο να καταρτήσει και να συμφωνήσει να ψηφίσει έναν κατώτατο μισθό. Αυτό όμως το οποίο μπορούμε να κάνουμε ε, για, ε, για τους πολίτες Ευρωπαϊκής Ενώσεως είναι εάν αυτοί δεν έχουν πρόσβαση εις ε, τις υπηρεσίες υγείας ε, της Ευρωπαϊκής Ενώσεως ή τις, ε, τις υπηρεσίες παιδείας και δικαιοσύνης και αυτά είναι στοιχεία που καθορίζουν την φτώχεια οπότε αποδεικνύεται <clears throat> ότι υπάρχει παραβίαση των θεμελιωδών δικαιωμάτων Πρέπει λοιπόν να εξασφαλίζει κανείς έναν κατώτατο μισθό, πρόσβαση στην παιδεία και πρόσβαση στην υγεία και την δικαιοσύνη για να ξεκαθαρίσουμε αν κάποιος βρίσκεται στο επίπεδο της φτώχειας ή όχι. Από εκεί και πέρα το επίπεδο ακριβώς του κατωτάτου μισθού δεν είναι τόσο σημαντικό και δεν είναι εύκολο να καθοριστεί διότι υπάρχουν ορισμένες χώρες όπου οι ε, χώρες δεν μπορούν ε, να ξεχωρίσουν τον κατώτατο μισθό από ε, αυτό το επίπεδο. Θέλω λοιπόν να σας ευχαριστήσω για όλες τις τροπολογίες και ελπίζω ότι και η αρμόδια επιτροπή θα δεχθεί αυτήν την έκθεση. Ευχαριστώ κυρία Ζαμπόρσκα. Αυτό ήταν το τελευταίο θέμα της ημερησίας διατάξεώς μας. Έχουμε περιθώριο για προθεσμίες μέχρι τις 15 Ιουλίου στις 12 το μεσημέρι. Δεν είναι πολύ καιρό ακόμη στη διάθεσή μας, αλλά υπήρχε μία ακόμη πιο στενή προθεσμία και θα ψηφιστεί 15 Σεπτεμβρίου. Ευχαριστώ για τη συνεδρίαση. Αύριο θα ξαναβρεθούμε ή στις 9 η ώρα το πρωί και αν τα καταφέρουμε θα μπορέσουμε να έχουμε την ευκαιρία κάποια στιγμή ε, να ευχηθούμε αλλήλεις καλές διακοπές. Η κυρία Ζαμπόσκα όμως φεύγει ήδη και τώρα θέλω να της ευχηθώ ένα ευχάριστο και χαλαρό καλοκαίρι. Θέλω να ευχαριστήσω και τους διερμηνείς και σας ζητώ συγγνώμη που ε, σήμερα ε, ε, ίσως τα μπέρδεψα σε ορισμένα σημεία. Πρέπει ιδίω να μην φοράω ακουστικά όταν μιλάω. Ευχαριστώ. Yeah.